Να ξεκινήσουμε. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των συντονιστών, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να έρθετε σε επαφή με τους συντονιστές σας ο καφής. Λοιπόν, για την ημερήσια διάταξη, συνάδελφοι. Αύριο στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έγκριση της γνωμοδότησης για την ε, πρόταση διαγραφής των διατάξεων του κανονισμού 1760-2000 σχετικά με την προαιρετική επισήμανση του βόηου κρέατος. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση ε, τροποποιημένη η οποία δεν ελήφθη υπόψη ε, κατά την εκπόνηση της γνωμοδότησης αλλά ούτε και κατά την κατάθεση των τροπολογιών. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τις 8 Μαΐου για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής και να ε, καθορίσουμε νέα προθεσμία για τροπολογίες 25 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι η πρόταση της Επιτροπής είναι η παριθμόν κομ 2012-162 και αν συμφωνείτε με την πρόταση αυτή θα ήθελα να ζητήσω και από την αρμόδια επί ουσίας Επιτροπή να αναβάλει και αυτή την ψηφοφορία. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις λοιπόν εγκρίνεται η τροποποιημένη μερίσια διάταξη. Να σας ενημερώσω επίσης αγαπητοί συνάδελφοι ε, ότι όπως γνωρίζετε από 1η ε, Απριλίου στα πλαίσια της διαδικασίας προσχώρησης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν παρατηρητής από το Κροατικό Κοινοβούλιο στη συνεδριά της Επιτροπής μας. Στην Επιτροπή μας λοιπόν έχουμε τον ε, συνάδελφο Μπόρο Γκρούμπιζιτ, τον οποίο και χαιρετώ. Νάτος εδώ. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Γκρούμπιτσης θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις μας και χαίρομαι ιδιαίτερα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον καλωσορίζω. Επίσης, στην Επιτροπή Γεωργίας έχουμε και ένα νέο αναπληρωτή από πλευράς Φιλανδίας, τον κύριο Πέτρη Σαρβάμα, τον οποίο επίσης καλωσορίζω. Ευχαριστούμε λοιπόν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε απευθείας στο σημείο 3 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 19ης και της 20ης Μαρτίου του 2012. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, τα πρακτικά εγκρίνονται. Και για σήμερα, όπως συνήθως, ε, η συνεδρία της Επιτροπής μας ε, μεταδίδεται μέσω web streaming ζωντανά στο διαδίκτυο. Σημείο 5. Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στα πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο εισηγητής, ο Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος, Να περάσουμε λοιπόν στο πιο σημαντικό σημείο της σημερινής συνεδρίασης, τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, κυρίως για το θέμα των άμεσων πληρωμών. Πρόκειται για ένα από τα βασικά ε, μεταξύ των τεσσάρων ζητημάτων και ίσως και το ένα από τα πιο δύσκολα και το πιο διαφιλομηνικούμενο. Είχαμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις και τώρα ο συγκητής θα μας παρουσιάσει τις βασικές θέσεις της, ε, γνω, τους και πριν δώσω το λόγο στο Λουίς, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βάσει χρονοδιαγράμματος θα παρουσιαστούν οι τέσσερι εκθέσεις στη συνεδρίαση τη Επιτροπής μας του Ιουνίου και κατόπιν η προθεσμία για την ε, κατάθεση των τροπολογιών θα είναι εντός του Ιουλίου. Τώρα, Λουίς, έχει το λόγο και κατόπιν θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τους τελευταίους τέσσερις με πέντε μήνες προσπαθήσαμε να έχουμε όσο δυνατό περισσότερες επαφές και ανταλλαγές απόψεων για το θέμα αυτό και εγώ πολύ περισσότερες ε, και όσοι συζητήσει για το θέμα αυτό. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς συναδέλφους, με πολλές οργανώσεις και συνεταιρισμούς γεωργών, πολλές οργανώσεις ε, για το περιβάλλον, με μέλη της κυβέρνησης, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης και έχω διαμορφώσει μια γνώμη σήμερα για τα πιο επίμαχα σημεία και για τα αλλά τα πιο συνενετικά σημεία που θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα όμως να σας ε, ε, εκφράσω την ε, απόλυτη διαθεσιμότητά μου και την προθυμία μου να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Με ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει σε μια στεναρή και συνεκτική άποψη κάτι που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική μα ισχύ απέναντι στο Συμβούλιο του επόμενου μήνε. Γι' αυτό και οι προτάσει που θα καταθέσω δεν είναι αποκλειστικά δικέ μου προτάσει, αλλά είναι προτάσει που κατά τη γνώμη μου μπορούν να συγκεντρώσουν ε, ω το δυνατό μεγαλύτερη πλειοψηφία. Θα ήθελα να ανατρέξω εν συντομία τα πιο νευραλγικά σημεία της έκθεσης. Καταρχήν, το πολύ δύσκολο θέμα της ανακατανομής. Όλοι συμφωνούμε ότι κάποιο είδους ανακατανομή θα πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί κάπως η άδικη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά κράτη-μέλη για τις ε, πληρωμές ανά εκτάριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της και εγώ θα καταθέσω μία εναλλακτική πρόταση. Μία εναλλακτική πρόταση που κατά τη γνώμη μου είναι πιο δίκαιη, απλούστερη και πιο κατάλληλη στο πολιτικό, οικονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο που ζούμε. Οπότε, τα κράτη-μέλη που είναι σε δυσμενή θέση, με την πρότασή μου θα βελτιώσουν κάπως την κατάστασή τους. Δεν θα ήθελα κανένα κράτος μέλος να μείνει κάτω από το 65% του κοινοτικού μέσου όρου. Και θα επιδιώξουμε μία σύγκληση, όχι για το 90% όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για 100%. Βέβαια, δεν θα είναι δυνατό όλοι να φτάσουν στο 90%, αλλά θα προτείνω σταδιακή αύξηση, πολύ μεγαλύτερη ε, για αυτούς που βρίσκονται στη χαμηλότερη πλευρά και ε, πιο αργή για όσους βρίσκονται πολύ κοντά στο μεσόρο. Και αυτός, αυτή η προσπάθεια ανακατανομής θα αντισταθμιστεί από τα κράτη-μέλη που έχουν μεγαλύτερη αναλογία δικαιούνται περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα του πρώτου πυλώνα. Όσα δηλαδή κράτη-μέλη έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, θα πρέπει αντίστοιχα να συμβάλλουν στην ανακατανομή. Κάτι που προϋποθέτει προσπάθειες μεγάλες από τα κράτη-μέλη που ξεπερνούν τον κοινοτικό μεσόρο. Και επαναλαμβάνω, κατά αναλογία. Φυσικά αυτή η λύση έχει κόστος, λίγο μεγαλύτερο από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επαναλαμβάνω αυτή η πρόταση ανακατανομής είναι πολύ πιο ε, μετριοπαθή σε σχέση με την ιδεώδη κατάσταση, αλλά με δεδομένη την κατάσταση είναι αυτή που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ε, πλειοψηφία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το greening, το πρασίνισμα της γεωργίας, οι προτάσεις που θα καταθέσω που δεν έχουν ακόμη αποκρισταλωθεί. Είμαι ανοιχτό, όπω σα είπα, στι προτάσει σα και στις υποδείξεις. Για το greening θα πρότεινα τα εξή. Καταρχήν, διαχωρισμός της βασικής πληρωμής από την πληρωμή για το greening. Θεωρώ ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η βασική πληρωμή ε, έχει την οικοαιρεσιμότητα, ενώ η συμπληρωματική πληρωμή του πρασινίσματος θα πρέπει να καταβάλλεται εφόσον τηρούνται οι όροι του greening. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες κυρώσεις για ε, μη συμμόρφωση, για παραβίαση. Αυτό όμως θα καθοριστεί από τον οριζόντιο κανονισμό για τον οποίο συγκεκριτής είναι ο κύριος Λαβία. Επίσης θέλουμε να διευκολύνουμε την χρήση των διαφόρων κριτηρίων ώστε ε, να επικεντρωθούμε στην εντατική γεωργία που προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον. Θα ήθελα λοιπόν τα μέτρα του πρασινίσματος, τα μέτρα του greening να ισχύσουν, να εφαρμοστούν με τρόπο που δεν θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικός. Επίσης θα ήθελα να πλουστευτούν κάπως τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στην περίπτωση του Ecological Focus Area, αλλά και στην περίπτωση της ε, διαφοροποίησης των καλλιεργειών, να εφαρμόζεται στις ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις άνω των τριών εκταρίων. Καλή αυτή η λύση, γιατί μιλούμε για μικρές ε, καλλιέργειες, όπου η πιθανότητα να κατηγορηθούν η γεωργή για μη συμμόρφωση είναι πολύ μεγάλη. και αυτό θα έλεγα αυτά τα δύο μέτρα να εφαρμοστούν κυρίως για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, άνω των 20 εκτάριων. Και σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταξύ 3 και 20 εκταρίων θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφοροποίηση μόνο μεταξύ δύο καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τα Ecological Focus Area, τις περιοχές ε, οικολογικής σημασίας, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια ενάυσματα στους γεωργούς που έχουν, κάποια, ε, έχουν ε, συνεχείς ζώνες οικολογικής προστασίας, ώστε να δημιουργήσουμε κάποιους διαδρόμους. Από τη στιγμή δηλαδή που μία εκμετάλλευση δέται με τη γειτονική, ε, θα πρέπει η απέτηση να είναι του, τάξη του 5 και όχι του 7%. Θα δημιουργήσουμε έτσι κάποιους οικολογικούς διαδρόμους. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικαιούχων αυτών των μέτρων, συμπεριλαμβάνοντας και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, που από άποψη οικολογικών πλεονεκτημάτων είναι ακόμη σημαντικότερα από τα μέτρα του, πρασιν, του που, και είναι αντίστοιχα με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία. Δηλαδή τα κράτη-μέλη ε, που έχουν γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα που είναι πιο απαιτητικά από τα μέτρα του greening, ε, η επιφάνεια που υπόκειται στα μέτρα αυτά θα πρέπει αυτόματα να θεωρείται ως ε, επιφάνεια που περιλαμβάνεται στα μέτρα greening, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιολογική γεωργία και τις εκμεταλλεύσεις που ε, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 2000. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα προστασίας του εδάφους, όπως οι, οι μόνιμες βοσκοτοπές, τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει να, να διαβρύνονται και σε άλλες μόνιμες καλλιέργειες, στο μέτρο που εφαρμόζονται γεωπονικές ε, πρακτικές προστασίας του εδάφους, της αναβάθμισης του εδάφους, δηλαδή ε, της διασφάλισης ε, χλώης στο έδαφος, εκεί που υπάρχουν ε, οι καλλιέργειες όπως είναι στις αμπελοϊνικές, στις απορροκυπευτικές, στις ελαιοκαλλιέργειες. Πρόκειται για μόνιμες καλλιέργειες που θα πρέπει να έχουν ένα επίπεδο προστασία του εδάφους αντίστοιχο με αυτό που ισχύει για τις μόνιμες χορτονομές. Νομίζω ότι στο greening, στο πρασίνισμα μπορούμε να περιλάβουμε πολύ περισσότερους γεωργούς από, αυτό, αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με απλούστερο τρόπο, γιατί οι τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς ελέγχου και εκεί που προτείνονται κάποιες διορθώσεις ε, της επιφάνειας ε, θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε τη γραφειοκρατία και ε, να περιορίσουμε κάπως, να ενισχύσουμε κάπως μάλλον την ελεκτική μας προσπάθεια. Και άλλε προτάσει θα μπορούσα να καταθέσω, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εσωτερική σύγκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη η ε, ενισχύσει ανεκτάριο να είναι ίσες για, ε, για όλους τους γεωργούς. Παρόλο που υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών στα ίδια το κράτος μέλος. Εγώ προτιμώ να υπάρχει ένα φάσμα ε, όταν μιλούμε για ποσοστό κάτω και πάνω από το μέσο όρο στο ίδιο κράτος μέλος, ώστε για να μην φέρουμε τους γεωργούς αντιμέτωπους μεταξύ τους ή τις περιφέρειες ενός κράτους μέλους σε αντιπαράθεση. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα τόσο μεγάλο εύρος ε, μεταξύ ε, του κράτους που, δέχεται, που λαμβάνει τις περισσότερες ενισχύσεις ανεκτάριο και αυτού που λαμβάνει τις λιγότερες ενισχύσεις ανεκτάριο και ε, αντίθετα εντός του ίδιου κράτους μέλους απαιτεί απόλυτη σύγκληση. Είναι τεράστια αντίφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα άλλο πολύ επίμαχο ζήτημα αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον ορισμό αυτό. Θεωρώ ότι ο ορισμός του ενεργού γεωργού θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός, αλλά να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους και ταυτόχρονα να καθοριστεί ένας αρνητικός κατάλογος επιφανειών, εκτάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τις άμεσες πληρωμές, γιατί σε αυτές δεν ασκείται καμία γεωργική δραστηριότητα. Για παράδειγμα αεροδρόμια, γήπεδα γκολφ, να έχουμε μία λίστα, έναν αρνητικό κατάλογο ε, επιφανειών που μέχρι στιγμής λάμβαναν παρόλο που δεν εκτελούνταν εκεί γεωργικέ εργασίε, αυτέ πια επιφάνειε να, εκ, να εξαιρούνται από τη δυνατότητα. Επίση, η μεταφορά μεταξύ των πυλώνων. Είμαι υπέρ της μεταφοράς αυτής μεταξύ των πυλώνων. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μερικές χώρες που έχουν μια κακή κατάσταση στον πρώτο πυλώνα και κάπως καλύτερη στο δεύτερο, να μπορέσουν να μεταφέρουν από το δεύτερο στον πρώτο. Αλλά θα πρέπει αυτές οι μεταφορές να περιορίζονται όσο γίνεται. Αλλά να μπορούμε να επιτρέπουμε κάποιες μεταφορές και από τον πρώτο προς το δεύτερο πυλώνα. Από αυτή την άποψη η πρόταση είναι καλή και θα μπορούσε να διατηρηθεί ως γενικός κανόνας το 10% από τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι για τα κράτη-μέλη που έχουν ένα πολύ ισχυρό πρώτο πυλώνα και έναν σχεδόν ανύπαρκτο δεύτερο πυλώνα. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ενάυσματα για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, ίσως με ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα, γιατί είναι μόνο 25% ο προϋπολογισμός του δεύτερου πυλώνα σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ και φυσικά αυτοί οι μηχανισμοί να προσαρμοστούν ανάλογα με το βάρος που έχει ο κάθε πυλώνα σε κάθε χώρα δεδομένων των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν και να είναι σημαντικές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους νέους Γιώργους, εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει υποχρεωτική αυτή η διάταξη και στο, στον, στην τόπα πληρωμή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία συμφωνώ για το θέμα της γύρασης του γεωργικού πληθυσμού είναι πολύ οξύ σε όλη την Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτή η top-up πληρωμή θα πρέπει να καθοριστεί με όριο επιφάνειας ίσο για όλους και όχι όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη μέση επιφάνεια της εκμετάλλευσης, η εκμετάλλευσης σε κάθε χώρα. Νομίζω ότι είναι ε, παράλογο ένας γεωργός που έχει 50 εκτάρια στη Ρουμανία να έχει τόπα μέχρι 6 εκτάρια που είναι ο μέσος όρος στη Ρουμανία και ένας γεωργός της Τσεχίας για παράδειγμα να μπορεί να λαμβάνει μέχρι 90 εκτάρια γιατί η, η μέση έκταση για τη γεωργική εκμετάλλευση στη Τσεχία είναι 90 εκτάρια. Νομίζω ότι η διαστάση μια γεωργική εκμετάλλευση σε μια χώρα δεν έχει καμία σχέση με το μέσο όρο των εκμεταλλεύσεων στη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό το κριτήριο λοιπόν, αν εφαρμοστεί, πραγματικά θα μας οδηγήσει σε πολύ γελία και παράλογα αποτελέσματα. Τέλος, ό,τι αφορά τη διατήρηση των συνδεδεμένων πληρωμών, μια διεκδίκηση ορισμένων χωρών μελών, θα πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη σοφροσύνη αυτό το μέτρο, αλλά να κρατήσουμε διαφυλάξουμε αυτή τη δυνατότητα, ώστε να μην ε, εξαφανιστούν ε, οι ορικέ δραστηριότητε τελείω από ορισμένε περιοχές. Να προβλέψουμε δηλαδή μία μεταβατική περίοδο. Και ένα άλλο επίμαγο θέμα είναι το ζήτημα του κάπινγκ και αυτό υπάρχουν πολύ αντιφατικές απόψεις. Θα ήθελα να πω ότι εγώ προσωπικά και η ομάδα μου είμαστε υπέρ ε, της φθήνουσας πορείας των ενισχύσεων και θα πρέπει να δούμε και το όριο, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος, αν είναι η καλύτερη μέθοδος αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουμε μία ευθύνουσα πορεία ανάλογα με τον αριθμό των εκταρίων. Πάντως, η αρχή της, ε, του φθήνοντα χαρακτήρα και η μεταφορά στο δεύτερο πυλώνα για την καινοτομία ή όχι μόνο για την καινοτομία, αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να διασφαλιστεί. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να κρατήσουμε και τη θετική διάκριση υπέρ της απασχόλησης. Γιατί έχουμε το ζήτημα των ειδικών δαπανών και των ε, μισθωτών που θα μειώνονται και θα λαμβάνουν την υπόψη στον υπολογισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους μικροκαλλιεργητές, τους μικρο... μικρής εμβέλειος γεωργούς, σε πολλές χώρες έχουμε πολύ σημαντικό κλάδο της μικρής γεωργίας, ενώ σε άλλες χώρες είναι ανύπαρκτη η μικρή εμβέλεια γεωργίας, εγώ θα πρότεινα να τροποποιήσουμε κάπως αυτό το καθεστώς, να ενισχύσουμε τους μικροκαλλιεργητές αφενός, αφετέρου όμως ε, να θέσουμε το μέτρο ως προαιρετικό, για να μην υποχρεώσουμε χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα ε, αναγκαστικά να πρέπει να θεσπίσουν κάποιες ενισχύσεις. Και τέλος, Να πω πάλι κάτι για το greening, κάτι που ξέχασα προηγουμένως. Πιστεύω ότι στο μέτρο που ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιεί το 30% του, τρι... του πρώτου πυλώνα που προορίζονται για το greening, αυτό το κονδύλιο θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα στο δεύτερο πυλώνα για να ενισχυθούν τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Γιατί αν θέλουμε να περιλαμβάνουμε στο greening τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και να κάνω αυτό το σύνδεσμο στο δεύτερο πυλώνα, θα είναι, σημαντικό να προβλέψουμε τα απαραίτητα κονδύλια στο δεύτερο αυτό πυλώνα. Γι' αυτό και θα προτείνω όχι μόνο προτείνουμε ένα ελάχιστο ποσοστό για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, αλλά ταυτόχρονα προτείνω ενίσχυση του κονδυλίου με κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται για το greening του πρώτου πυλώνα. Αυτά, Αυτές είναι οι προκαταρκτικές μου ιδέες. Είμαι ανοιχτό όπως είπα, στη συζήτηση και διαλλακτικός. Περιμένω τις προτάσεις και όσες προτάσεις κρίνω πιο δίκαιες, απλούστερες και καλύτερες, φυσικά θα τις περιλάβω με μεγάλη ευχαρίστηση στην έκθεσή μου. Επαναλαμβάνω, στόχος μου είναι με πνεύμα συνεργάσιμο και διαλεκτικότητας να καταλήξουμε σε μια στεναρή θέση συνενετική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικές γιατί για τι ριζοσπαστικέ προτάσει, δεν νομίζω ότι θα συγκεντρώσουμε συμφωνία, γιατί για αυτέ απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Δεν νομίζω ότι θα συγκεντρωθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο για μια ριζοσπαστική πρόταση που δεν θα βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε με επικοδομητικό τρόπο να επιφέρουμε κάποιε βελτιώσει και κάποιε καινοτομίε στο αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για την προσοχή τους. Ε, ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα και σας κούρασα. Ευχαριστώ Λουίς. Ε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, επομένως ε, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει και η μεταξύ μας συζήτηση. Επισημαίνω και στον εισηγητή και στους κοιόδης εισηγητές ότι πρέπει να υπάρχει πολύ στενή συνεργασία διότι ε, η δύναμη της Επιτροπής μας θα είναι ανάλογη της ευρύτερης πλειοψηφίας που θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ευθύ εξ αρχής να είναι κοινέ κάποιες ευαισθησίες. Να ξεκινήσει η συζήτηση, είναι πάρα πολύ εγγεγραμμένη, να προσπαθήσουμε λοιπόν να διαχειριστούμε λίγο το χρόνο μας ε, όσο το δυνατόν καλύτερα, δύο-τρία λεπτά ο καθένας, ε, να ξεκινήσει από τον κατάλογο που έχει ετοιμάσει η γραμματεία, ο George Lyons και μετά ο Jim Nicholson. George. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καπουλά Σάντο για τη συνεργασία. μαζί με μένα και με άλλους σκιώδες συζητητές σε ό,τι αφορά τις ιδέες που αποτυπώνονται. Θα ήθελα να διατρέξω λίγο κάποια από τα θέματα τα οποία έθιξε και ο ίδιος. Να πω εξ αρχής ότι συνολικά η κατεύθυνση που έχει επιλέξει δεν με βρίσκει αντίθετο. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως εξακολουθεί να προσεγγίζει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρά να αποτυπώνει την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό εν γέννη θα περάσω σε λεπτομέρειες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναδιανομή και τη χρήση του 100% ως τον αντικειμενικό στόχο, αντί για το 80% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι λεπτομέρεια και δεν πρόκειται να είμαι επιθετικός, αλλά θα πρότεινα ότι οι χώρες εκείνες με το μεγαλύτερο όγκο θα πρέπει να είναι υπεύθυνε για τη συμβολή στην αναδιανομή αυτή. Να δούμε τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι από τη Γερμανία και από τη Γαλλία για το θέμα του πρασινίσματος, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μία από τις κριτικές που δεχτήκαμε ήταν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, είναι μία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη αυτή η θέση. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μία γκάμα μέτρων. Σε ό,τι αφορά τις ξεχωριστές θέσεις ε, των κρατών μελών σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά την ε, διάκριση από την πληρωμή, τη βασική πληρωμή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή θέση σας και θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε και να δούμε και ποιες θα είναι οι κυρώσεις. Και φυσικά θα πρέπει να κοιτάξουμε και πάλι τι έχετε να προτείνετε συγκεκριμένα για την γραφειοκρατία, αλλά νομίζω ότι γενικά ότι οτιδήποτε απλοποιεί την κατάσταση το καλωσορίζουμε. Μία πρόταση τώρα για τις περιοχές οικολογικής ε, επικέντρωσης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρόμους ε, λέτε και να μην έχει κάθε καλλιέργεια, κάθε εκμετάλλευση μια ε, περιοχή εκρανάπαυσης. Αυτό να το κοιτάξουμε. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που αφορά πάρα πολλές χώρες είναι οι πληρωμές από τις ε, η μετάβαση από τις ιστορικές πληρωμές στις ε, ε, πληρωμές ανά Ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας φαίνεται ότι έχει θέσει αυτό το στόχο των ελάχιστων και των ανώτατων ε, προϋποθέσεων για τους γεωργούς, για να υπάρχει μία εξίσωση σε ό,τι για παράδειγμα αφορά το 120% ε, σε σχέση με τις ε, μέσες πληρωμές κτλ. Είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά μήπως ε, δεν χρειάζονται κάποια κυριαρχία εθνική. Δεν αναφερθήκατε στο πόσο α, μεγάλες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν, για παράδειγμα, τεράστιες αλλαγές που θα συνεπάγεται το σύστημα αυτό για κάποιους γεωργούς και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε κατά πόσον αποτελεί ένα σωστό βήμα για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διαφορές ύψους 30-40%. Θεωρώ ότι θα πρέπει να περιοριστούμε γύρω στο 10%. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και την χρονική περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση. Δεν είμαι βέβαιος ότι το 2019 είναι η σωστή χρονική στιγμή για τα πιο πολλά άλλα ζητήματα. Για το κάπινγκ, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι για... θα είμαστε αντίθετοι, διαμετρικά αντίθετα, αντίθετοι σε ό,τι αφορά το κάπινγκ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι και πολλοί άλλοι θα είναι αντίθετοι για τα πράσινα κονδύλια, τα οποία, θα πρέπει, τα οποία τα χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να μεταφέρονται. Συμφωνώ. Συνολικά και ανακεφαλαιώνοντας. Είναι πάρα πολλοί οι τομείς στους οποίους ε, θα πρέπει να βρούμε συμφωνία και μπορούμε να βρούμε συμφωνία, αλλά Νομίζω ότι θα πρέπει η θέση του Κοινοβουλίου γενικά να είναι πολύ πιο ε, διακριτή σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριος ε, και μετά κύριο Λόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το ζήτημα η θέση του είναι πολύ ισορροπημένη και χαίρομαι που ε, ανέλαβε και πάλι, είναι πάλι επί το έρχον. Η πρώτη παρατηρήση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ό,τι και να γίνει μετά από το 2014 δεν θα πρέπει να είναι άλμα από τον κρεμό. Θα πρέπει να είναι μία οδός προς ένα χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια, όπου οι γεωργοί θα έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν για την αλλαγή. Ε, γιατί ναι μεν θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές αλλά όχι να τους ε, έχουμε και τις αλλαγές να κρέμονται ως δαμάκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους να υπάρχει χρόνος να προσαρμοστούν όσον αφορά το greening το μετριασμό των συνεπειών ε, του περιβάλλοντος συμφωνώ με τις θέσεις που υπάρχουν και από πλευράς μου θεωρώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και στην έκθεση, αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι γεωργοί επιτόπου. Δεν είμαι υπέρ ε, του ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό που προτείνεται και δεν θα πρέπει να βρίσκεται στον πυλόν αυτό για το greening. Ό,τι και να γίνει θα πρέπει να είναι απλουστευμένο και θα πρέπει να απλουστευτεί. Το πρόβλημα είναι ότι όταν λέμε ότι πρέπει να απλουστευτεί και η πρόταση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν είναι τίποτα απλό αυτή την πρόταση και δεν ξέρω πώς θα μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά χωρίς περισσότερη γραφειοκρατία και ε, περισσότερο άχθος για όλους. Και πολύ με ανησυχεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι γεωργοί θα δημιουργήσουν έναν συμπληρωματικό κατάλογο και από αυτό τον κατάλογο θα μπορούν να δράσουν και θα αλλάζει ο κατάλογος στα διάφορα κράτη-μέλη διότι ε, σίγουρα δεν ταιριάζουν σε όλους ε, όλα και θα πρέπει σε κάποια κράτη-μέλη να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας για να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, εγώ προσωπικώς θα ήθελα να αφαιρεθούν τελείως από το κείμενο αν πρέπει να γίνουν, ε, να υπάρχουν, θα πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς ε, στους οποίους ίσως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους περιβαλλοντικούς φορείς και εκεί η γεωργοί είναι ήδη δραστηριοποιημένοι σε αυτές τις δράσεις, αλλά δεν θα πρέπει να τις πληρώσουν δύο φορές οι γεωργοί τις περιοχές αυτές. Και όσον αφορά τώρα τις μόνιμες καλλιέργειες και τα μόνιμα βοσκοτόπια, Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ σαφείς ε, ως προς τις θέσεις μας και τι ακριβώς πρέπει να εννοεί ε, το συγκεκριμένο. Εγώ ξέρω πολλές γιες οι οποίες δεν έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί τους τελευταίους 12 μήνες, αλλά η πλειονότητα των περιοχών στις οποίες ε, περιέρχομαι εγώ, προέρχομαι εγώ είναι βοσκοτόπια και διατηρούνται ως μόνιμα βοσκοτόπια. Ξέρουμε λοιπόν πώς να το κάνουμε. Τώρα για το κάπινγκ, εγώ από πλευρά μου διαφωνώ με το κάπινγκ. και κάποια μέλη που έρχονται από τις νέες χώρες ε, γνωρίζουν πόσο δύσκολο θα είναι να το προσεγγίσουμε αυτό και εγώ το συνειδητοποιώ απολύτως και στην ομάδα μου και η πολιτική μου ομάδα το συνειδητοποιεί απολύτως. Θα γίνει μακρά συζήτηση από αυτού και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν θα φτάνουμε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, όταν και όποτε θα γίνουν. Πρέπει η λήψη αποφάσεων να γίνει από κάτω προς τα πάνω για να ξέρουμε πολύ καλά πώς έχει η κατάσταση επιτόπου. Όσον αφορά τώρα τους ε, ενεργούς γεωργούς, εγώ προσπάθησα να βρω κάποιον ο οποίος να το υποστηρίζει και ακόμα δεν έχω βρεθεί ε, ενώπιον κάποιου που, που μου είπε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογο ως αυτών που δεν επιτρέπονται. Δεν χρειαζόμαστε γήπεδα γκολφ, δεν χρειαζόμαστε ανοησίες. Θα πρέπει να είναι γέες οι οποίες χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν φτάσουμε ε, στον ορισμό του ενεργού γεωργού, τελικώς θα δημιουργήσουμε κάτι τόσο γραφειοκρατικό που θα δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό άχθος και θα είναι φιάλτης κατά την άποψή μου. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι αυτού ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρκετά ποσά στο δεύτερο πυλώνα για το θέμα αυτό και αυτό τους έχει δημιουργήσει αρκετές δυσκολίες. για να υπάρχει ένας πυλώνας ο οποίος θα είναι στη μορφή που αναμένει ο καθής και επισημαίνω λοιπόν ότι στον πυλώνα 2 χρειάζονται κάποια ε, περισσότερα κονδύλια για να εφαρμόσουμε όλες τις περιβαλλοντικές πολιτικές που χρειάζονται. Και να τελειώσω και με μια τελευταία παρατήρηση, η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Την περασμένη εβδομάδα το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ιδιαίτερα επικριτικό για το πακέτο της μεταρρύθμισης. Ε, είπαν ότι θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και θα είναι και προβληματικός προς τη διαχείριση. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι θα στοιχίζει 15% επιπλέον η διαχείριση αυτών των αλλαγών. Εγώ δεν ξέρω καμία κυβέρνηση πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που έχει το περιθώριο ή ελπίζει να έχει τη δυνατότητα να έχει ένα 15% δαπάνη επιπλέον για τη διαχείριση της γεωργικής της πολιτικής. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη δεν είναι εφικτό όσο έχει αυτή τη στιγμή να έχουμε μία αύξηση 15% επιπλέον στη γραφειοκρατία για τους γεωργούς. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το σημείο κλειδί Εάν δείτε αυτό το 15% είναι σημαντικά αυτά τα ποσά σε πάρα πολλές περιοχές και είναι σίγουρα χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή όταν έχουμε πει σε χώρες ότι πρέπει να γίνει δημοσιονομικός έλεγχος, πρέπει να μειώσουν τις δαπάνες τους και εμείς τώρα τους ζητάμε να έχουν επιπλέον κονδύλια για να διαχειριστούν αυτά τα θέματα. Ε, είμαι βέβαιο, βέβαια ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή για να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση και ελπίζω τελικώ και η Επιτροπή μας ε, ε, για την έκθεση αυτή αλλά και για όλε τι υπόλοιπε εκθέσει που αφορούν την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική να καταλήξουμε σε μία ισχυρή θέση ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο και, το Ευρωπαϊ... και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι σαφέ ότι θα είναι θετική η συνεισφορά μας. Τώρα, η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και όπω και οι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, όχι μόνο για την πολύ καλή παρουσίασή του εδώ πέρα σήμερα, αλλά και για τι συναντήσει ε, των τελευταίων εβδομάδων. Θα είμαι σύντομη και θεωρώ ότι ε, μία από τι δυσκολίε για την Επιτροπή μα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, λεπτομέρειε, αλλά είναι περιορισμένο ο χρόνο μα για την πρότασή σα για την αναδιανομή. Κινείται προ μία κατεύθυνση που ικανοποιεί κάποιους άλλους όχι. Για το θέμα λοιπόν αυτό θα είναι δύσκολο να πετύχουμε μια απόλυτα συμφωνία και ξέρω ότι οι, τα κράτη-μέλη δεν θα ικανοποιηθούν ούτε με την πρόταση αυτή. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Αλλά και επίσης εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης δυσκολίας του προϋπολογισμού και της χρηματοδότησης Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέμα των εκτελεστικών πράξεων και των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Θα χρειαστεί κάποιο ορισμό. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι σίγουρο ότι έχουμε τον έλεγχο των θεμάτων αυτών πριν τον ε, χάσουμε τον έλεγχο. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες των όσων προτείνονται για την, ε, τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Κανείς δεν συμφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ωστόσο θα πρέπει να κοιτάξουμε το συνδυασμό ενδεχόμενης αρνητικής λίστας και μπορεί να εξετάσουμε την, το άρθρο 28 του κανονισμού 73 του 2009, γιατί ο κανονισμός αυτός ήδη επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ορίσουν και να καταργήσουν κάποιου ορισμού σε ό,τι αφορά τι χειρουργικέ δραστηριότητε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτή που θα δώσει κάποια ευελιξία για το κάπινγκ των πληρωμών. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τα νούμερα, τα αριθμητικά στοιχεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, αν ε, μειώνουμε, αν μειώσουμε τους μισθού όπως προτείνεται, θα πρέπει να δούμε και το κόστος των συμβάσεων, των συμβασιούχων μάλλον των ε, αγροτών, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις, ανατίθεται σε, σε, μέσω σύμβαση σε κάποιους η συλλογή κάποιων καρπών, για παράδειγμα. Αυτά είναι, όλα αυτά είναι, αποτελούν κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη για να είμαστε δίκαιοι για την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων. Αυτό θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν τι τους ταιριάζει καλύτερα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα βρίσκεται σε μια νεκτική θέση. Το αφήνω λοιπόν στην παρούσα φάση το θέμα αυτό. Να κοιτάξουμε το θέμα του πρασινίσματος και της σύγκλησης. Τώρα, για την πρόταση για το πρασίνισμα, για το greening, αυτό που ήθελε στην έκθεση Desk Lion το Κοινοβούλιο είναι αυτό που αναφέρεται, ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι περίπλοκο το οποίο θα εφαρμόζεται χωρίς ε, περιττές γραφειοκρατίες. Είπατε όμως, Πρόεδρε, ότι αυτές είναι οι πιο δύσκολες ε, μεταρρυθμίσεις που έχουμε επεξεργαστεί ως τώρα. Αληθεύει αυτό. Καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι τα πλεονεκτήματα τροποποίησης των μέτρων κατά τον τρόπο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταστούν πιο πρακτικά σε επίπεδο γεωργού, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει οι ε, εναλλακτικές λύσεις που έχουν τα κράτη-μέλη να είναι πιο ποικίλε προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιο πολλές συναρκτικές λύσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ότι κάποια κρατημέλη δεν έχουν τέτοιες ε, ε, περιοχές οικολογικής, ε, οικολογικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία λίστα που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιλέξει για παράδειγμα δύο μέτρα για κάθε γεωργό, γιατί το τρέχον σύστημα επιβάλλει να χρησιμοποιηθούν και τα τρία αυτά μέτρα, το οποίο δεν είναι δίκαιο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τι προτείνουμε για τα μέτρα πρασινίσματος. Συμφωνώ με την ιδέα σας ότι πρόκειται, ιδέα σας ότι πρόκειται για ξεχωριστή πληρωμή και ο γεωργός δεν θα πρέπει να εξαναγκάζεται να εισέλθει στο καθεστώς αυτό να μην υπάρχει κύρωση σε περίπτωση που αποφασίσει να μην συμμετάσχει στις βασικές πληρωμές. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα για το πρασίνισμα, τα οποία όμως είναι υπερβολικά, αν θέλετε, λεπτομερή. Να κοιτάξουμε το θέμα της σύγκλησης, το οποίο συνδέεται με τα θέματα πρασινίσματος. Το ανέφερε και ο George Lyon, το θέμα της μεγάλη ε, διαφορά που υπάρχει. Αν πάρουμε το συν 40% που αναφέρεται στο άρθρο 22, μιλάμε για προσαρμογή 58%. Για κάποια κρατημέλη αυτό είναι αδύνατο. Νομίζω λοιπόν ότι την ιδέα της προσέγγισης που προτείνεται πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες φυσικά, αλλά ενδεχομένως να λειτουργήσει. Να μας πείτε επίσης κατά πόσον η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταργηθεί σε όλα τα κρατημέλη το σύστημα των δικαιωμάτων κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί ξέρω ότι τα παλαιά κρατημέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τα νέα κρατημέλη και αυτά τα κρατημέλη που έχουν ιστορικές πληρωμές. Και το ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ ε, σύνθετο και πολύ σύνθετο για τον ε, εισηγητή. Το βασικό όμως θέμα που θα αυξήσει το κόστος το, βασικό μάλλον είναι ότι θα αυξήσει το κόστος για τα κρατημέλη, γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα για το τι δικαιούται και τι πληρώμε δικαιούται ο καθένα. Ίσως λοιπόν θα χρειαστούν τροποποιήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θεωρώ ότι η σύγκληση είναι εξίσου πολιτικά ευαίσθητη όσο και το πρασίνισμα, ίσως και πιο πολύ. Γιατί όταν θα καταλάβουν οι γεωργοί πια ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις εκμεταλλεύσεις τους, θα είναι μεγάλη η αντίδραση και ίσως να πρέπει να προτείνουμε και μία ενδιάμεση αναθεώρηση, μία ανάλυση του αντίκτυπου του πρασενίσματος και της σύγκλησης όσο πλησιάζουμε και κινούμαστε προς το 2019. Μιλήσαμε για τα σχέδια του αγροτικού περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το παρόμοιο καθεστώ του με την βιολογική γεωργία. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που θα αποτυπώνουν την πρόταση αυτή που την είχαμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή. Για τις πληρωμές προς τους νεαρούς ε, γεωργούς. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σύστημα. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν και αποκλήσεις και απόψεων ακόμα και στην ειδική μου ομάδα και σε όλο το Κοινοβούλιο. Η πρόταση που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι θα λειτουργήσει για τους νεαρούς γεωργούς. Γι' αυτό λοιπόν θα βρούμε κάτι πιο πρακτικό. Χρειάζεται κάπως χτένισμα αυτή η πρόταση για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. για τη συνδεδεμένη στήριξη. Δεν ξέρουμε ποιο επίπεδο θα ήταν σωστό για το σχέδιο για τον μικρό γεωργό. Μπορεί να μην φαίνεται κατάλληλο αυτό ως πρόταση, αλλά ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μια ε, εναλλακτική λύση στα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, ίσω μακρηγόρησε και ξεπέρασε το χρόνο που μου είχατε δώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω πολλέ λεπτομέρειε ακόμα να αναφέρω. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ντόρφαν και μετά ο Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Ε, κάποια λίγα σημεία θα ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά το πρασένισμα που ανέφερε ο εισηγητής. Θεωρώ ότι είναι λογικό και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα κατώτατο όριο, το οποίο θεωρώ είναι τα 20 εκτάρια. Οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα μεταρρύθμιση του περιβάλλοντο δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν με περαιτέρω μέτρα πρασινίσματο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Και επίσης ότι θεωρώ ότι είναι καλό και αποτυπώνει τις φιλοδοξίες ε, για την γεωργία όταν τα χρήματα αυτά δεν ε, χρησιμοποιούνται να μεταφέρονται στο δεύτερο πυλώνα. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις για την ιστορική σύγκληση. Νομίζω ότι η ιδέα για να ρίσουμε ένα ποσοστό για την ιστορική σύγκληση είναι σωστή και λογική. Αρκεί να μιλάμε για το σύνολο ενός κράτους και όχι για συγκεκριμένες περιφέρειες. Και αυτό ισχύει για χώρες που υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ της μίας περιοχής και της άλλης περιοχής. Εγώ αναφέρομαι πάντα στην Ιταλία. όπου η αναλογία είναι ένας προς δέκα, μία περιοχή προς δέκα. Και αυτή η δυσαναλογία είναι πολύ μεγαλύτερη από τις δυσαναλογίες που υπάρχουν μεταξύ χωρών. Αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το επιλύσουμε. Δεν συμφωνώ επίσης να ορίζει κάθε χώρα ξεχωριστά την ορισμό του ενεργού γεωργού. Γιατί θα καταλήξουμε στο ίδιο πρόβλημα ε, που έχουμε αυτή τη στιγμή με τις μειονεκτικές περιοχές που μας το ε, επισημαίνει κάθε φορά το ελεκτικό συνέδριο Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μεν ε, η αρχή της επικουρικότητας, αλλά νομίζω ότι ο βασικός κανόνας θα πρέπει να μπει στον κανονισμό και όχι να ορίζεται από κάθε κράτος μέλος μόνο του για τους μικρούς γεωργούς. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής. και θεωρώ ότι το ανώτατο όριο δεν θα πρέπει να ορίζεται από τα χρήματα που παίρνουν από τον πρώτο πυλώνα, αλλά από την επιφάνεια τους, από την έκταση τους. Αυτό θα ήταν πολύ πιο απλό στην προσμέτρηση, γιατί τα χρήματα ε, μπορεί να διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο. Ένα τελευταίο ζήτημα. Μία ερώτηση προς τον εισηγητή. Δεν είπατε τίποτα για τις μειονεκτούσες περιοχές. Σε ό,τι αφορά τον να υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Ευχαριστώ τον Έρμπερτ, τον Ζωζέ Μποβέ. Και μετά ο κύριος Ολένιτσακ. Ευχαριστώ. Όντως, ε, συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τον εισηγητή και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Όπως ε, ενδιαφέρουσα είναι και αυτή η απογευματινή συζήτηση που έχουμε, γιατί καταδεικνύει και τα σημεία σύγκλησης, αλλά και την ανάγκη να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να περιοριστούμε σε ορισμένα θέματα. Σε ό,τι αφορά καταρχήν τη σύγκληση των κρατών μελών. Αυτό το θέμα το συζήτησα με τον εισηγητή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να θεσπίσουμε ένα όριο διάρκειας. Όταν βλέπουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φτάνουμε και πέρα το 2028 μερικές φορές. Νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε μία ημερομηνία, να θεσπίσουμε ένα χρονικό όριο για να οριοθετήσουμε κάπως α, τις προτάσεις. Αλλιώς θα είναι πολύ άδικη η κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι στις βαλτικές χώρες και σε άλλες χώρες που μπήκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι εύκολο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ενεργών γεωργών. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες, είναι πολύ λογικό αυτό που μας είπε. Να ορίσουμε όχι με θετικό τρόπο τι εστί ενεργός γεωργός, αλλά με αρνητικό τρόπο, δηλαδή τι δεν αποτελεί ενεργό γεωργό. Και από τη στιγμή που θα το ορίσουμε κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία που να μην εμπίπτουν στο θέμα του ενέργου Γιώργου. Είπαμε για το εισόδημα. 90% του εισοδήματο ε, να μην προέρχεται από τη γεωργία. Σε τέτοια περίπτωση δεν είναι κάποιο που το 90% του εισοδήματό προέρχεται από μη γεωργικέ δραστηριότητε να χαρακτηρίζεται γεωργό, ούτε μπορεί να ε, δικαιούται ενισχύσει. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα, μια σαφή άποψη. Σε ό,τι αφορά το κάπινγκ το, τον θέσπιση ανώτατων ορίων και την φθήνουσα μείωση των ενισχύσεων. Τη σταδιακή μείωση των ενισχύσεων, συγγνώμη. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι υπερβολικοί οι περιορισμοί και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αρκετή. Άλλοι θεωρούν ότι το ανώτατο όριο είναι υπερβολικά ψηλό και εγώ θα προτιμούσα να μειωθεί αυτό στα 100.000 ευρώ. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάποια ανακατανομή των κονδυλίων, θα πρέπει ο περιορισμός να είναι αποτελεσματικός για να δημιουργηθεί μια ε, μάζα κονδύλιων. Και μάλιστα δεν θα πρέπει όσοι έχουν αποφεληθεί από εδώ μέχρι τώρα ρωτόρια να τροφοδοτήσουν ε, την ανακατανομή. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε εσωτερικά την ανακατανομή μεταξύ των Γεωργών. Νομίζω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Σε ό,τι αφορά το κλίμα και τη γεωργία και το περιβάλλον, το greening δηλαδή. Και εκεί θα πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους. Να δούμε ποια είναι η μελλοντική γεωργία που θέλουμε. Δηλαδή, να μην περιοριστούμε σε μόνο, μόνο σε τεχνικά μέτρα, αλλά να πούμε ότι μας ενδιαφέρει ε, μια βιώσιμη γεωργία, ένα βιώσιμο γεωργικό σύστημα για τη δεδομένη των κλιματικών αλλαγών, της θέρμας του πλανήτη, της ποιότητας του εδάφους, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι φτάνουμε, οδεύουμε προς μια μετάλλαξη του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου. Δεν έχουμε μόνο θέμα προσαρμογής δηλαδή των μέτρων, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο μοντέλο θέλουμε για τη γεωργία μας. Τι, τι είδους γεωργία θέλουμε να υποστηρίξουμε και να διαμορφώσουμε στο μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι σε ορισμένα θέματα δεν θα μας ακολουθήσει η πλειοψηφία, αλλά το λέω ότι θα πρέπει σταδιακά να εφαρμόσουμε το greening, να να ξεκινήσουμε από το 25% και στο 2020 να φτάσουμε στο 50%. Ένα προοδευτικό σταδιακό σύστημα ώστε το, το μερίδιο της ε, ενίσχυσης προς τους α, ε, ε, γεωργούς για το greening να φτάσει σταδιακά μέχρι το 50%. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό το μήνυμα για την τροποποίηση του γεωργικού συστήματος που επιδιώκουμε. Ένα άλλο σημείο σχετικό, το συζητήσαμε και όλα, το θέμα της διαφοροποίησης. Δεν συμφωνώ με τον όρο αυτό, γιατί διαφοροποίηση, ε, όταν έχουμε μία καλλιέργεια 70% ε, δεν νομίζω ότι μιλούμε για πραγματική διαφοροποίηση. Σε ό,τι αφορά τις πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης, ε, λέει η Επιτροπή ότι αν περιλάβουμε εδώ και την παραγωγή της σόγιας ή πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης, ε, θα μας κατηγορήσουν στον ΠΟΕ για να Έχουμε λοιπόν μια μετάλλαξη προς αυτονομία σε πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης. Δεν θα πρέπει να ενταχθούμε σε μια λογική διαφοροποίησης, αλλά σε μια λογική αμυ, Οπότε θα μείνει χωρίς επιχειρήματα και ο ΠΟΕ, γιατί θα έχουμε τελείως διαφορετικό μοντέλο. Αμυψησπορά λοιπόν, εναλλαγή των καλλιεργειών, κάθε ένα-δύο χρόνια, ε, με σταδιακή εισαγωγή των, των καλλιεργειών ε, ψυχανθών και για παραγωγή ε, πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης. Ό,τι αφορά τις μικρές ε, καλλιέργειες. Και εκεί χρειαζόμαστε ένα όραμα. Τι θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις για να τις βοηθήσουμε σταδιακά να εξαφανιστούν ή θέλουμε ε, να διασφαλίσουμε την παρουσία της στο, στη γεωργία. Οπότε η στήριξη αυτών των μικρών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να στηρίξει και δίκτυα μεταποίησης, διανομής... Και εκεί μπορούμε να το συνδυάσουμε το δεύτερο πυλώνα για να, για να δημιουργήσουμε υποδομές επιτόπου και να δώσουμε εργαλεία στις μικρές εκμεταλλεύσεις για να επιβιώσουν. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό της μικρής εκμετάλλευσης του μικροαγροκτήματος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ορισμένες περιπτώσεις η επιφάνεια, η έκταση, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον κύκλο εργασιών, που είναι σημαντικό κριτήριο για να καθοριστεί ε, κατά πόσο μια εκμετάλλευση είναι μικρή ή μεγάλη. Γιατί μια γεωργική εκμετάλλευση δύο εκταρίων ε, στην Καμπανία δεν είναι μικρή εκμετάλλευση. Μια ε, εκμετάλλευση στην Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία για κτηνοτροφία, αυτή όντω εμπίπτει στον ορισμό τη μικρή εκμετάλλευση. Ένα συνδυασμό κριτηρίων λοιπόν για να καταλήξουμε στον ορισμό τη μικρή εκμετάλλευση. Και εγώ πάντως ε, θα ήθελα να πρωτοστατήσει το Κοινοβούλιο στη συζήτηση αυτή και να μην αφήσει μόνο τους το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί στο Συμβούλιο θα δημιουργηθούν αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών μελών. Εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καθορίσει την ακολουθητέα πορεία, να ενισχύσει την παρουσία του και ευχαριστούμε θερμά τον εισηγητή. Ευχαριστώ Ζωζέ. Το λόγο έχει ο κύριος Ολέινιτσακ. Ε, και θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους ομίλητες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λουίς Καπόλα Σάντος για το έργο του που βάζει κάποια τάξη στη συζήτηση και ταυτόχρονα διαπιστώνουμε από τη συζήτηση πόσο δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας και πόσο λίγος χρόνος μας έχει μείνει ώστε να ετοιμάσουμε για τους γεωργούς εν ώψη του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου μια καλύτερη γεωργική πολιτική. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το ύψος των ε, πληρωμών σύγκλησης, το κυρίως θέμα. Και εγώ είμαι υπέρ της ισότητας ε, των πληρωμών για όλους τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια κακή λύση και αυτό που προτείνει ο Λουίς οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε αν είναι και η λύση του Λουίς επαρκής. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να εφαρμόσουμε ίσες ε, ισότιμες πληρωμές. Και νομίζω ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η άποψη καλό θα ήταν να πριτανεύσει. Επίσης ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτήσει όλες αυτές οι λύσεις να εφαρμοστούν πανευρωπαϊκά. Όλες αυτές οι προδιαγραφές δηλαδή να ισχύουν και να δεσμεύουν όλα τα κράτη-μέλη. Και να μην ε, αφήσουμε πολλά πράγματα στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, γιατί έτσι δεν θα έχουμε κοινή γεωργική πολιτική, αλλά γεωργικές πολιτικές που θα έχουν εθνικό χαρακτήρα. Το ίδιο ισχύει και για το greening, για το πρασίνισμα. Κάπως πιο ελαστικές προτάσεις ουσιαστικά ε, διαψεύδουν τις προσδοκίες των γεωργών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε στα 20 εκτάρια, αυτό είναι, να είναι το σωστό επίπεδο. Νομίζω επίσης ότι αυτή η λύση θα πρέπει να ισχύει για όλους τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως η πρόταση αυτή των 20 εκταρίων είναι μια σωστή πρόταση προς τη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα του ενεργού γεωργού και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να οριστεί πανευρωπαϊκά. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε σε κάθε κράτος μέλος. Θέλουμε κοινό μοντέλο. Η μέση γεωργία ε, ή μάλλον ε, πόσα εισοδήματα προέρχονται από ελληνικές δραστηριότητες. Πολύ σημαντικό. Και από τη στιγμή που οι ενισχύσεις δεν εξυπηρετούν τη γεωργία αλλά άλλες δραστηριότητες, αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες μεταφοράς μεταξύ των πυλώνων. Επίσης, ε, κάτι που δεν διευκρινίζεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι θα γίνει δηλαδή με τα ε, κονδύλια το 30% που δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν για το, για greening μπορούν να περάσουν στο δεύτερο πυλώνα. Πιστεύω ότι ναι. Είναι πολύ δίκαιη αυτή η πρόταση και ε, οι, οικονομ... οι εκμεταλλεύσεις που σήμερα και στο μέλλον θέλουν να είναι οικολογικές, να μην πρέπει επιπλέον να έχουν και γραφειοκρατικό άχθος για να ε, φτάσουν στο 30% του greening. Γιατί είναι προφανές ότι πληρούν όλα τα κριτήρια. Γιατί αυτός ο ορισμός είναι πολύ πιο δύσκολος. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θεμελιώδες ζήτημα. Εμείς θα πρέπει σε κάθε αλλαγή να εξετάσουμε και το κόστος της και τη γραφειοκρατία που επιφέρει. Δηλαδή, αν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα τμήμα της πρότασης προϋποθέτει γραφειοκρατικό άχθος, ενίσχυση του γραφειοκρατικού άχθους και δυσχεραίνει τους γεωργούς, του απαιτεί να αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο ε, για διατυπώσεις, για γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι για τη γεωργική εκμετάλλευση, τέτοιου είδους ε, λύσεις θα πρέπει να τις αποκλείουμε. Δεν θέλουμε λύσεις που να επιτείνουν το γραφειοκρατικό άχθος, γιατί αυτό δεν θα το καταλάβουν ούτε οι γεωργοί. Οι γεωργοί θέλουν να είναι στη γη τους, δεν θέλουν να συμπληρώνουν χαρτιά συνέχεια. Ούτε εκείνη η γνώμη θα αντιληφθεί πώ είναι δυνατόν να εγκρίνουμε μια πρόταση με τόσο έντονο γραφειοκρατικό άκθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ολόνιτσε. Ε, και τώρα η Ελίζα Μπεθ και μετά ο κύριος Καλινόσκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον εισηγητή για την επικοδομητική ε, εργασία και για την καλή συνεργασία εν γέννη. Θα ήθελα σήμερα να καταλαβαίνω πορτογαλικά γιατί ειλικρινά η απλοποίηση των προτάσεων για το πρασίνισμα όπως μας παρουσίασε ο εισηγητής σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν σαφής. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα με την πρόταση σε ό,τι αφορά το greening. Κυρίως σε ό,τι αφορά θέματα διοικητικά και ε, θέματα ελέγχου. Να πω ότι αν το ελεκτικό συνέδριο τώρα ήδη από το πρώτο βήμα μας επισημαίνει πόσο ακριβή θα καταστεί η γεωργική πολιτική και ξέρουμε ε, ότι ο θετικός αντίκτυπος στη γεωργία δεν έχει σχέση με το κόστος που συνεπάγεται. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν να σκεφτούμε κατά πόσον αυτός ο λογαριασμός ε, αυτός ε, είναι λογικός. Γιατί και οι γεωργοί θα έχουν λιγότερα χρηματοδοτικά μέσα στη διάθεσή τους στην περίπτωση αυτή. Και θα ήθελα να ξέρω επίσης ε, τι σκοπεύει να κάνει ο εισηγητής ε, ό,τι αφορά τις ε, περιοχές οικολογικής επικέντρωσης. Και να πω ότι θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα θα είναι στον τομέα του ελέγχου. Ένα παράδειγμα από την Αυστρία, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ απλό σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκτάσεων, αλλά στην πράξη έχουμε τεράστια προβλήματα κάθε χρόνο σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των πραγματικών εκτάσεων. Κρύω τον κόδωνα λοιπόν του κινδύνου και σας ε, επιστήνω την, την προσοχή σας. Και σε θέματα εφαρμογής θεωρώ ότι θα υπάρχουν προβλήματα, γιατί θεωρώ ότι η βιώσιμη γεωργία είναι πιο σωστή προσέγγιση από το να αφαιρεθούν συγκεκριμένες εκτάσεις και μετά πάλι να υπάρχει η υποχρέωση ελέγχου. Θεωρώ λοιπόν καλύτερο είναι να υπάρχει μια γενική προσέγγιση. Επίσης, ε, πολύ ε, ενδιαφέρον ε, Βρίσκω αυτό που προτείνει ο εισηγητή για τη μεταφορά του 30% στον δεύτερο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν τα μέτρα αυτά για το πρασίνισμα. Αλλά θα ήθελα και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην έκθεση να μην εξαντλούνται σε περίπτωση που δεν εξαντλούνται τα ε, μέσα αυτά, γιατί κάποια μπορεί να μην μπορούν, να μην θέλουν να τα εξαντλήσουν αυτά στο πρώτο πυλώνα, να μπορούν τουλάχιστον να το κάνουν μέσω του δεύτερου πυλώνα. Να παρατηρήσω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα μεταξύ των γεωργών σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή δεδομένων και το μέτρο λιτότητας που λαμβάνονται σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι μεγάλη λοιπόν η αβεβαιότητα και γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να υπάρχει μια σαφή τοποθέτηση της Επιτροπής ε, Γεωργίας και να αναλάβουμε τις ευθύνε μας στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας για την προσπάθεια που έκανε να δημιουργήσει μία άποψη μεταξύ των αντιπαρατεθειμένων χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, ίσως η αντιπαράθεση δεν είναι σωστός όρος, αλλά πραγματικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των, ε, της γεωργίας στη γεωργία των κρατών μελών και αυτό είναι πολύ δύσκολο για τον εισηγητή, καθίστα πολύ δύσκολο για τον εισηγητή την ανέβρεση λύσεων. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί και το, συγχαίρω γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το greening, έχουμε σημαντικές απαιτήσει για τους γεωργούς στα πλαίσια ε, του, της ανάγκης λήψης υπόψη του περιβάλλοντος και έχουμε ενιαίες απαιτήσει, αλλά οι αντισταθμίσεις, οι επιβραβεύσεις δεν είναι ισότιμες. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 30% από τα εθνικά κονδύλια. Δηλαδή, αντί να, να προσπαθήσουμε να εξισώσουμε τις υποχρεώσεις, εμβαθύνουμε και οξύνουμε ακόμη περισσότερο τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, γιατί δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες. Εμείς προτείνουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα με ίσες και αντισταθμίσεις. Είμαι υπέρ της, του ορίου που προτείνεται για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Νομίζω ότι η πρόταση του εισηγητού οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, όλα τα πλονεκτήματα του greening ε, να μην τα λαμβάνουμε μόνο από μια καλλιέργεια. Ε, αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό και με, την, ε, με τον ορισμό. Ποια είναι η πράσινη γεωργία, ποια είναι η πράσινη ε, γεωργική εκμετάλλευση. Είναι αυτή που εφαρμόζει και περιβαλλοντικά προγράμματα ή προγράμματα στα πλαίσια του Natura 2000. Θα πρέπει να δούμε και τον ορισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Επίσης, ε, τι λήψη υπόψη της οικολογικής διάστασης. Έχουμε πολλές μεγάλες διαφορές στην Ευρώπη. Και όσο μεγαλύτερο κατακαιρματισμό στις γεωργίες υπάρχει, όσο περί, περίπλοκη είναι η δομή, τόσο μικρότερα είναι και τα αγροτεμάχια. Εμείς ε, έχουμε σε 20 εκτάρια 30-40 εκμεταλλεύσει πολλέ φορές. Αν θέλουμε ε, να έχουμε αποσύνδεση όχι σε κάθε αγροτεμάχιο αλλά σε κάθε δύο, θα έχουμε περίπου 10 εκατομμύρια μικρά, πολύ μικρά αγροτεμάχια ε, με το ecological ε, ε, focus, αυτή την οικολογική εστίαση. Πώς είναι δυνατόν να ελέγξουμε ένα τέτοιο σύστημα, αποκλείεται. Επίσης το θέμα των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης που ανέφερε ο κ. Μποβέ. Νομίζω ότι η επιφάνεια για την καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων καλλιεργιών φυτικής πρωτεϊνών φοιτική προέλευση. θα πρέπει να ε, περιληφθούν αυτές οι εκτάσεις στην οικολογική καλλιέργεια. Άλλωστε, τέτοιου είδου καλλιέργειε βελτιώνουν και αναβαθμίζουν και το έδαφο. Οπότε θα πρέπει να επιβραβευτεί η χρήση, η επέκταση τέτοιων καλλιεργειών ψυχαθών και πρωτεϊνών φυτική προέλευση. Η Ελίζαπεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή μα. Και εγώ θα ήθελα να μπορώ να αντιληφθώ κάποιες ε, γλωσσικές, αν θέλετε, λεπτομέρειες για να καταλάβω και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί σίγουρα το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σύνθετο για το πρασινίσμα, για τον πρωτοπυλώνα. Αυτό με αναπασχολεί ιδιότερα και η διάκριση με το δεύτερο πυλώνα με τέτοιο τρόπο που να μην ε, αποβείς βάρος των συμβατικών, αν θέλετε, Γεωργούς. Δεν κατάλαβα αρκετά α, ε, τις λεπτομέρειες, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε για το 30% για το πρασίνισμα. Το 7% των ε, εκταλέσεων θα προσθεθεί επιπλέον και 30% είναι 7% τι θα γίνει με τις μειονεκτικές περιοχές στην όλη ιστορία αυτή. Τι θα γίνει με τα υφιστάμενα προγράμματα για την ε, γεωργική εκμετάλλευση και αυτό που αναφέρθηκε το Natura 2000. Όλα αυτά τα οποία δηλαδή ήδη υπάρχουν. Πώς μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στον τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη και προκειμένου να ληφθούν υπόψη και το σύνολο των εκμεταλλεύσεων για τον ορισμό των διαδρόμων και αυτή η βιολογική εφαρμογή. Κατάλαβα ότι και αυτό θα πρέπει να αποτελεί σημείο εστίαση. Κάποια στιγμή, όχι απαραίτητο σήμερα, να μου πείτε πώ ακριβώς. Μία παρατηρήση να κάνω για την αναδιανομή. Νομίζω και αυτό το λέω συνειδητά ως Γερμανίδα βουλευτής. Θεωρώ λοιπόν ότι τα τελευταία, την τελευταία αγροτική μεταρρύθμιση την πήραμε πολύ στα σοβαρά και στη Γερμανία ολοκληρώσαμε τις ε, περιφερειακές πληρωμές χωρίς ε, να υπάρχει αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ιστορικές πληρωμές. Τώρα τι ακούω, ότι για πολλά κρατημέλη, για πολλούς γεωργούς σε κάποια κρατημέλη, η κατάσταση δυσχεραίνεται εξαιρετικά. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε συνολικά με πλειοψηφία το θέμα αυτό και θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει το πιο δύσκολο ζήτημα και νομίζω ότι πολύ βασικό είναι και αυτό το η τάξη, αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση που τη βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά από κάθε παράγραφο. Θα πρέπει να ορίσουμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά σημεία κλειδί για μας και θα πρέπει να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κοιτάξτε εδώ πέρα δεν μπορείτε να μας ε, υποσκελίσετε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα ζητήματα αυτά. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Σιγητά. Ευχαριστούμε την Ελίζα Μπεθιέγκελ. Πράγματι το θέμα των πράξεων ε, εξουσιοδότηση από την συνθήκη της Λισαβόνας θα περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Μάρτιν Όσλιν και μετά η Μπρίτα Ρέινς. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή καταρχάς γιατί νομίζω έκανε συζητήσεις με όλες τις ομάδες και συχνά προσπάθησε να συμπεριλάβει προτάσεις ε, των άλλων ομάδων. Δεν μπορούμε φυσικά με 2.000 ε, τροπολογίες να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα. Για αυτά τα οποία ακούσαμε από τον εισηγητή σήμερα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σίγουρα θα πρέπει να συζητηθούν και συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή ότι δεν επαρκεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αναδιανομή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει δικαιοσύνη στην ε, ε, ΚΑΠ. Για να επανέλθουμε όμως ε, στον πυρήνα της μεταρρύθμισης που νομίζω έγκυται στο πρασίνισμα, στο greening. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να τηρήσουμε την αξιοπιστία μας σε ό,τι αφορά και το Κοινοβούλιο και το βρικινό. Η εντύπωσή μου είναι η εξή ότι το όλο greening, το όλο πρασίνισμα, θεωρείται ότι δεν είναι πλέον τόσο απαραίτητο. Θεωρείται ότι είναι, τι να πω, ένα μικρό παράρτημα. Αν ξεκινήσουμε να ορίσουμε ένα βασικό πόσο πληρωμών και δεν το συνδέσουμε με το πρασίνισμα, διευκολύνουμε όλους όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν και παίρνουν τη βασική πληρωμή και πολύ απλά δεν συμμετέχουν στη συνέχεια. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Δεν μπορούμε να απαλλάξουμε όλη τη γεωργία από την ευθύνη της και να πούμε ότι όσοι θέλουν να το κάνουν, όσοι δεν θέλουν να το κάνουν. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό. Και αν βάλουμε κάποια εμπόδια, όπως τα 20 εκτάρια για παράδειγμα, σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται να πετύχουμε οποιοδήποτε άξιο σημείο το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα για το πρασίνισμα και τι θα βγούμε θα πούμε στους πολίτες μετά. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το αξιοσημείο το αποτέλεσμα που θα έχουμε πετύχει με το πρασίνισμα. Δεν νομίζω ότι στατιστικά θα έχουμε οτιδήποτε να παρουσιάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάποια σημεία να συζητήσουμε για το greening και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θεωρώ ότι ούτε καν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκεί. Θέλουμε λοιπόν Αν θέλουμε να υπάρχουν, για παράδειγμα, τέτοιε πληρωμέ, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρία είδη, για παράδειγμα, ε, καλλιεργειών. Και θεωρώ ότι να δούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται με τις ε, τιμές της ε, σόγιας, για παράδειγμα όπου 80% για παράδειγμα εισάγεται, ενώ παράλληλα καταραίουν οι τιμές του γάλακτος. Δεν μπορούμε τέτοιες διαφορές να τις αποδεχόμαστε γενικά. Όλα θα πρέπει, αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την κοινή αγροτική πολιτική για το τι είναι ενεργός γεωργός. Θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση ο εισήγητης. Η λύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ γραφειοκρατική. Και η αρνητική λίστα νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να ορίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Ποιος να παίρνει τα χρήματα και ποιος όχι. Και ότι κάποιοι απλά δεν έχουν δικαίωμα για τέτοιες πληρωμές από τον κοινό Κορβανά. Συμφωνώ επίσης με τον Σοζέ Μποβέ Νομίζω ότι με, τις, ε, το σημερινό μοντέλο του κάπινγκ δεν έχουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Ή θα πρέπει να ξεκινήσουμε πιο νωρίς με το κάπινγκ γιατί θα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στο, κοινοβούλιο, στο, στο κοινό γιατί αποδεχόμαστε ακόμα ε, την υποστήριξη των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Θα έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να δικαιολογήσουμε τα μέτρα αυτά και αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθήσουμε νομίζω από πλευράς του Κοινοβουλίου Δεν θα πρέπει τελικά όμω να κάνουμε τόσο πολλέ υποχωρήσει έναντι του, του Συμβουλίου που τελικά να μην παραμείνει τίποτα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειαζόμαστε τη γεωργική μεταρρύθμιση και ότι θα πρέπει από κοινού να την εφαρμόσουμε και ότι θα πρέπει τελικά ο φορολογούμενος να καταλάβει πιο πολλά από την μεταρρύθμιση από την τελευταία φορά. Και θα πρέπει λοιπόν ο εισηγητής να τηρήσει και να εμείνει στις θέσεις του και σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με το Συμβούλιο, γιατί στην αγροτική μεταρρύθμιση αποτελούμε ένα σημαντικό παράγοντα για τον καθορισμό της νέας κατεύθυνσης. και δεν θα πρέπει να κάνουμε υπερβολικούς συμβιβασμού από τόσο πρώιμη φάση. Αυτό είναι το δικαίωμα που έχουμε ως Κοινοβούλιο και νομίζω ότι μπορούμε να το περάσουμε και πάρα πολύ σωστά προς τα έξω, προς, το, προς τους πολίτες. Grazie. Martin, adesso Britta Reimers. Ευχαριστώ. Τώρα η Μπρίτα Ρέιμοντς και μετά ο κύριος Η κυρία Το τελευταίο καιρό αμφιβάλλω για το κατά πόσο ξέρουμε τι κάνουμε εδώ στην αγροτική πολιτική. Έχουμε όλο και πιο πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική κρίση και ε, δέχονται πιέσει οι εθνικοί προπολογισμοί. Έχουμε κυβερνητική κρίση σε πολλές χώρες και η πίεση αυτή, αν δεν μειωθεί, θα είναι τεράστια και η πίεση και σε ό,τι αφορά τον αγροτικό προϋπολογισμό. Και τώρα να καθόμαστε και σκεφτόμαστε πόσο περίπλοκα ε, μπορούμε να κάνουμε την αναδιανομή, όλα αυτά δεν πρόκειται να αντέξουν. Βλέπω πώς προσπαθείτε να βρείτε συμβιβασμούς μεταξύ των διαφορετικών γραμμών, αλλά εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο ξέρουμε τι κάνουμε πραγματικά γιατί βλέπω ότι απομακρυνόμαστε από τον πραγματικό μας στόχο, από το να θεωρούμε δηλαδή τους αγρότες ως ανεξάρτητους επαγγελματίε. Κινούμαστε προς μια κατεύθυνση όλο και πιο πολύ προς ε, διαμόρφωση πολιτικών στρατοπέδων ε, για ιδεολογικούς ε, σκοπούς πάντα κινούμαστε προς την κατεύθυνση να προδιαγράφουμε ε, στους γεωργούς το τι θα καλλιεργούν, πώς θα το καλλιεργούν, γιατί και πάλι και με το greening θα προδιαγράφουμε πώς θα καλλιεργούν οι αγρότες. Δεν τους αφήνουμε ελευθερία. Εμείς θέλαμε προς την αντίθετη κατεύθυνση να κινηθούμε. Και τώρα και πάλι ξεκινάμε τις παρεμβάσεις στην αγορά αυτή. Σκοπός θα έπρεπε να είναι μακροπρόθεσμα να βγούμε από το καθεστώς των άμεσων πληρωμών προκειμένου να είναι πραγματικά ελεύθερος επιχειρηματίας ο Γεωργός. Αλλά στην παρούσα φάση δεν ε, βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αν το ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι τουλάχιστον να το κάνουμε σωστά, πιο έντονα, για να μην υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό απογοήτευσης μεταξύ των γεωργών. Κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και πολίτης δεν δέχεται όλη αυτή την αύξηση της γραφειοκρατίας να την πληρώσει σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα της Γεωργίας. Νομίζω ότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν έπρεπε να είναι στον πρώτο πυλώνα το πρασίνισμα. Θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στο δεύτερο πυλώνα και να συνοδεύεται από ένα σωστό περιβαλλοντικό πρόγραμμα με την αναλογή χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα είχαμε πετύχει πιο πολλά σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Το θέμα όμω είναι ότι δεν έχει γίνει αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπω έχει και εγώ πολύ φοβάμαι ότι όσο πιο πολύ το συζητάμε τόσο πιο πολύ περιπλοκό θα γίνει το ζήτημα αυτό. Και όλο και πιο πολύ παρεμβαίνουμε στα προσωπικά δεδομένα των ε, γεωργών. Τώρα θέλουμε να μας δώσουν την ε, τιμή, το κόστος. Αυτό κάνουμε με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναρωτιέμαι. Όπως σας είπα, ε, η μεγάλη απογοήτευση θα οδηγήσει πολλούς γεωργούς το να αποχωρήσουν από το και να αφήσουν τις δραστηριότητε τους. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Μπρίτα. Και τώρα η κυρία Καλνιέτε και μετά η κυρία Ρανς Καρσία κατόπιν έχουμε τους κύριους Γιάρνταν, Τέρνε, Ντες, Σαβά και Βατσεβόσκη και κατόπιν θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα για τις μειονεκτικές περιοχές, ενώ το σημείο ε, για τη μεταφορά των ζώων αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρία του κυρίου Βατσεβόσκη. Κύριε Καρνιέτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τακούλα Σάντος που θέλει να βελτιώσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να συμφωνήσω και με όλους εκείνους όσοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να εξευρεθεί συμφωνία. Μιλάμε για άμεσες πληρωμές και για αναδιανομή. αν κάποια κράτη τα οποία λαμβάνουν πιο, πολύ, πιο πολλά από ότι άλλα κράτη δεν είναι πολιτικά διατεθειμένα να κάνουν ένα βήμα προς τα πίσω. Κοιτάξτε, αυτό είναι καταρχάς πολιτική απόφαση. Εκ παραλλήλου θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι αυτή η ανισόρροπη διανομή των άμεσων πληρωμών ε, προέκυψε ιστορικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί σε μία, αν θέλετε, άνηση κατάσταση, σε, μια, σε έναν άνισο ανταγωνισμό. Και για να μην έχουμε την εντύπωση ότι τα κράτη της Βαλτικής ζητούν ε, κάτι ειδικό για τον εαυτό τους, να σας πω ότι έχουν την κάθε πρόθεση να αναλάβουν το 100% των άμεσων πληρωμών. Αλλά αυτό να ισχύει για όλους. Το θέμα είναι λοιπόν να μην υπάρχουν πλέον τέτοιες διαφορές προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική και στο παγκόσμιο προσκήνιο η γεωργία. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι στα κράτη της Βαλτικής λαμβάνουμε τις πιο μικρές πληρωμές και παράλληλα καλούμαστε να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις και όλους τους όρους που εκπληρώνουν και τα υπόλοιπα κρατημέλη, ακόμα και Κίνα, τα οποία λαμβάνουν τετραπλάσια, εξαπλάσια ποσά από ό,τι εμείς. Και οι άμεσες πληρωμές συνδέονται με τις βασικές τιμές, με την έκταση. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι η εκτάσεις μας εξαγοράζονται από άλλους πολίτες, από άλλους γεωργούς, από άλλα κράτη-μέλη που δεν μπορούν, γεωργούς που δεν μπορούν να αγοράσουν γη στη δική τους χώρα. Σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Λετωνία, είναι πολύ χαμηλές οι τιμές για την ε, σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις. Τέλος, να πω ότι τα κράτη της Βαλτικής παρακολουθούν εντελεχώς τα ζητήματα τα οποία συζητούμε εδώ σε ό,τι αφορά την υποστήριξη προς τους νέους ε, γεωργούς. Το επόμενο θέμα τώρα για το πρασίνισμα. Είμαστε πραγματικά ε, πολύ εξελιγμένα κράτη σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα αυτό και μας φαίνεται ότι είναι υπερβολικό το 7%. Το ίδιο ισχύει και το ορισμό του ενεργού γεωργού. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας. αγανάκτη, η κοινή γνώμη για τους γεωργούς εκείνους που λαμβάνουν ε, ποσά υποστήριξης, χωρίς όμως να είναι ενεργή. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ενός συμβιβασμού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στη γεωργία χρειάζονται συμβιβασμοί προκειμένου όλοι να είναι τελικά κερδισμένοι και να μην ε, βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα είναι επιζήμια για όλους. Και επίση θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τι ειδήσει για τον, τη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή. Σα ευχαριστώ. Αλλά σας θέρμα παρακαλώ, ρίχνετε και μια ματιά στο ρολόι, στο χρονόμετρο, για να μην ξεπερνάτε κατά πολύ το χρόνο σας. Λυπάμαι που σας το υπενθυμίζω, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ γενναιόδοροι με το χρόνο. Κύριε Ραντ Καρσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι επιτέλους δημιούργησε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου για να συζητήσει ε, τα θέματα τα αμπελουενικά, τα οποία ήταν τα πιο σημαντικά το τελευταίο καιρό και επίσης ε, να απορρίψω την ε, ε κατάργηση των ποσοστώσεων για το ζάχαρη, διότι υπάρχουν κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα ε, η αγορά αυτή των ζαχαρότευτλων που είναι πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια. Τώρα, για την έκθεση του κυρίου Καπούλα Σάντος, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δέξουμε ιδιαίτερη προσοχή στο κατά πόσον θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να διατηρήσουμε, συγγνώμη, άμεσες ενισχύσεις ε, σε περιοχές ε, οικολογικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν κάποια μέτρα, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει διπλή χρηματοδότηση και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί εδώ και να το μελετήσουμε προσεκτική. Όσον αφορά το greening τώρα, αυτή την ιδέα που προτείνεται. Πραγματικά εμένα μου φαίνεται βαρβαδρότητα να έχουμε αυτό το 20% για το greening και παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο είναι ε, βοήθεια θεωρητικά είναι, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπως ο κτηνοτροφικός τομέας που δεν έχουν καμία βοήθεια από ουθενάλλου. Και επίσης ήταν ο Επίτροπος εκεί στην Ισπανία αυτές τις μέρες και εξέτασε τα θέματα του, του ελαιολάδου. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε το greening σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο greening ε, για μια χώρα ε, της Βόρειας Ευρώπης με μια χώρα ε, η οποία είναι καθαρά αγροτική όπως είναι οι, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ε, ενδιαφέρονται τα μας προτείνει ο εισηγητή για τον ενεργό γεωργό και το ενδιαφέρον είναι ότι θεωρείται ενεργό γεωργό, αυτό που έχει κάποια παραγωγική δραστηριότητα. Βέβαια δεν πρέπει να είναι η μοναδική του δραστηριότητα, αλλά άμα δημιουργεί θέση εργασία και δημιουργεί η πλούτο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ω ενεργή γεωργή ανεξάρτητα από το μέγεθο τη εκμετάλλευση. Γιατί μία μικρή εκμετάλλευση όπου κάποιο αυτό απασχολείται έχει το, κάθε, το ίδιο δικαίωμα να θεωρείται ενεργή παραγωγή, ακόμα και αν ε, στη συγκρίνουμε μια εκμετάλλευση όπου, στην οποία εργάζονται, απασχολούνται 50 άτομα. Ε, πάντα σε αυτή την περίπτωση τους θεωρούμε όλους ενεργούς γεωργούς. Και τέλος, Αναφερόμαστε πάντα στα ιστορικά κριτήρια, αλλά θα πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε και πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει και κάποιε ιδιαιτερότητε για ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν τομείς, όπω για παράδειγμα το μέας του ρυζιού και του ελαιολάδου, που είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να έχουν σημαντικέ εξαιρεσει, διότι θα έχουν άμεσες επιπτώσεις με την εφαρμογή των μέτρων και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και επίσης να σας πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιου τομεί όπω την εντατική εκτινοτροφία που δεν έχει εδαφική βάση. Αυτή η αποσύνδεση επίση ε, είναι επιπλέον ποσόστοση η οποία γίνεται σε αυτή την περίπτωση και σε κάποιε περιπτώσει δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με κάποιου τομεί όπω είναι αυτή, όπω και με όλου του υπόλοιπου και να μην υπάρχει διάκριση για κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ ε, καλή δύναμη στον εισηγητή, κάνει πολύ καλή δουλειά και να συνεχίσει. Ευχαριστώ. δεν ξέρω πόσα λεπτά θα χρειαστεί ο εισηγητής ε, για να απαντήσει. Ο κύριος Γιάρ και μετά ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή γιατί δεν είναι εύκολο το έργο του. Θα προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε όσο γίνεται να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Τέσσερα σημεία έχω γράψει, τέσσερις παρατηρήσεις για τις άμεσες πληρωμές πρώτον. Συμφωνώ. Θα είμαστε πιο γρήγοροι από ό,τι πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σας παρακαλώ δύο πράγματα. Καταρχάς, παρακαλώ να λεφτούν υπόψη οι διαφορές μέσα στους τα κρατημέλη. Πολλές φορές αναφέρθηκαν αυτό. Ξέρω ένα γεωργό που δεν λαμβάνει άμεσες πληρωμές και έχω μάθει ότι οι διαφορές εντός των κρατών μελών είναι πιο μεγάλες από ό,τι μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές στο εσωτερικό των κρατών μελών. Το ανέφερε και η κυρία Γέγκλε. Θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και σε ό,τι αφορά το health check. Ένα δεύτερο πρόβλημα. Συζητούσαμε μια αντιπροσωπεία από τα κράτη της Βαλτικής που μου ανέφεραν ότι μεγάλο τμήμα των εκτάσεων δεν είναι καταχωρισμένο γιατί τη στιγμή της ε, ε, προσχώρησης ε, ήταν εκμετάλλευση ρωσική. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των άμεσων πληρωμών, αλλά το πρόβλημα είναι και οι καταχωρισμένες εκτάσεις. Θα ήταν δηλαδή πολύ ε, κακό να επηρεάσει έτσι η ρωσική κατοχή του, την, τη σημερινή ε, πληρωμή της, ε, των χωρών αυτών για την μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει, για παράδειγμα, ορισμός του ενεργού γεωργού να σας προειδοποιήσω, γιατί οποιαδήποτε διευκρίνηση θα ε, προκαλέσει ένα γραφειοκρατικό ε, κυκλώνα και πολύ το φοβάμαι αυτό. Γιατί αυτά που θέλουμε να πετύχουμε δεν θα τα πετύχουμε. Γιατί θεωρώ ότι αν η βασίλισσα της Αγγλίας ε, πάρει ένα καλό λογιστή θα μπορέσει να της αποδείξει ότι είναι και αυτή η ενεργός γεωργός άμα θέλει. Προσέχετε λοιπόν για το πρασίνισμα. Η πρόταση που συχνά ακούσαμε για τη σύνδεση με το δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να μη συνδέεται με όρους για το greening. Ε, εγώ και η συνάδελφος Γέγκλε σπάνια συμφωνούμε. Αλλά κοιτάξτε, άμα συμφωνούμε μία φορά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή αυτή η πρόταση. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τρίτο σημείο για το cupping. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Είμαι κατά του μέτρου αυτού. Επειδή επί του προεχομένου δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Θα πρέπει να χαιρόμαστε αν οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις θεωρούν ότι ανήκουν σε κάποια οικογένεια. Γιατί αυτό που προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι είναι ε, ο σχηματισμός βιομηχανικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Θα προκύψει ένα βιομηχανικό ένας βιομηχανικός κλάδος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να το αποφύγω αυτό σε ό,τι αφορά το κάπινγκ. Θα πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μία ακρόαση. Έχουμε κοιτάξει τι έγινε με τον καπνό, με το γάλα, με τη ζάχαρη καταλαβαίνω ότι υπάρχει τάση στην Επιτροπή να παρατείνουμε τα μέτρα. Ίσως θα έπρεπε να το κοιτάξουμε ξεχωριστά το θέμα αυτό, γιατί Ναι, μεν είναι αντίθετα προ τα συστήματα τα μέτρα αυτά, αλλά υπάρχουν και λόγοι για του οποίου θα μπορούσαμε να τα διατηρήσουμε. Και πάλι κάθε επιτυχία εύχομαι προ τον εισηγητή. Ελπίζω να είναι επιτυχή η έκθεσή του και να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των μελών στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ το λόγο κύριο Ντε. Όχι, ο κύριο Νταντά πρώτα και μετά ο κύριο Ντε. Άντε κύριε Ντες πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λουίς Καπούλα Σάντος και για τις συζητήσεις που εξηγεί μαζί μας και θα ήθελα να πω συνοψίζοντας το εξής παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συζήτηση όλων των ε, ζητημάτων αυτών η πρόταση του Καπούλα Σάντος λίγο πολύ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πιο πολύ από ότι σε σχέση με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι' αυτό λοιπόν θα τη βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόταση αυτή με βεβαίως κάποια σημεία τώρα τα οποία θα ήθελα να υποστηρίξω θα ήθελα να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ των βασικών πληρωμών και των πράσινων πληρωμών. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσέγγιση την οποία μπορούμε να συζητήσουμε και για το μέγεθο των επιχειρήσεων, των εκμεταλλεύσεων από 3 σε 20 εκτάρια. Θεωρώ ότι και αυτό είναι πολύ καλή πρόταση. Επίσης, τι άλλο θα πρέπει να συζητήσουμε, τα μέτρα για το πρασίνισμα. Και εδώ είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι απόψεις μας, όπως φάνηκε και είναι και πάρα πολύ διαφορετική η κατάσταση κατά κράτο μέλο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεωρώ ότι οδηγεί σε πιο πολύ γραφειοκρατικό άχθος και θεωρώ ότι δεν το... αυτό είναι το μοναδικό που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεδομένης και της κατάστασης των ε, λιτότητας που επικρατεί στα κράτη-μέλη, δεν είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μια κατάσταση στα κράτη-μέλη όπου η Γεωργία θα έχει 20% πιο πολύ γραφειοκρατία. Δεν πρέπει να το δεχτούν αυτό οι Γεωργοί. Θα πρέπει να ξέρουμε τι κονδύλια έχουμε στη διάθεσή μας και τι μπορούμε να ζητάμε από τους γεωργούς. Εγώ Πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή μου έχουμε τιμές που εκτοξεύονται στα ύψη, τριπλάσιες, τετραπλάσια. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το να πούμε ότι χρειάζεται αγρανάπαυση 7% των εκτάσεων είναι απαράδεκτο. Ε, για παράδειγμα, ένας ε, γεωργό στην περιοχή μου ε, έχει 20% της εκμετάλλευσης που ε, καλλιεργεί μόνο στην ιδιοκτησία του και αν τον υποστηρίξουμε, αν τον υποχρεώσουμε να βγάλει εκτός παραγωγής το 7% πολύ απλά ε, οι τιμές ενοικίασης των εκτάσεων θα αυξηθούν στα ύψη. Θα πρέπει, για παράδειγμα, υπολογίσαμε για το συγκεκριμένο Γιώργο να πληρώνει 8.000 ευρώ περισσότερο ποσό σε ό,τι αφορά την εκμίσθωση. Τέτοιε προτάσει πραγματικά δεν μπορούν ε, να αποτελέσουν το μέλλον της γεωργίας. Είπε ο αδελφο Σέραντς ότι τα μέτρα για το πρασίνισμα από την Φιλανδία μέχρι τη Σικελία, από την Πορτογαλία μέχρι τη Βουλγαρία δεν μπορούν να είναι τα ίδια, γιατί η Ευρώπη διαφέρει, αν θέλετε έχει είναι πολύ μεγάλη πολυμορφία που παρουσιάζει και τα κράτη-μέλη διαφέρουν. 20% των χρηματοδοτικών των ε, αγροτικών πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μέτρα λογικά για το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε. Τελευταίο σημείο για να μην ε, μακρηγορώ, ο ενεργός γεωργός. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με χιούμορ σε κάποιες περιπτώσεις, ε, Πρόεδρε. Θα ήταν χρήσιμο ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει μία πρόταση για το τι είναι ο ενεργός υπάλληλος. Ίσως στην περίπτωση αυτή βάσει τη πρόταση που θα μα υποβάλουν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι είναι ο ενεργός γεωργός για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να μας κάνουν μια εκτίμηση για να καταλάβουμε. Τελευταίο ζήτημα για να διανομή μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό των κρατών μελών θα πρέπει να γίνει πιο δίκαια από ό,τι προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον εισηγητή προκειμένου τελικά να βρούμε μια καλή λύση για τους γεωργούς μας. Σας ευχαριστώ κύριος Ντάντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις διευκρινήσεις που έκανε και τα στοιχεία που πρόσθεσε στη συζήτηση. Το, το greening, το πρασίνισμα δεν είναι κακή πρόταση, αλλά ο τρόπος που προτείνεται να εφαρμοστεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ακατάλληλος και ε, δυσνόητος και για τους ε, γεωργούς. Ε, όπως φαίνεται και αυτό που είπε ο κύριος Αλμπέρ, ο νέος γεωργός θα πρέπει να συνεχίζει να λαμβάνει τις ενισχύσεις της ΚΑΠ για τα 7 εκτάρια που θα αφιερώνει στη βιοπικιλότητα. Αλλιώς θα επιβαρυνθεί ε, και θα στερηθεί ένα μεγάλο τμήμα των ενισχύσεων. Ο εισηγητής μας πρότεινε κάποια διαφοροποίηση και διευκρίνησε κάπως ε, τα δεδομένα της συζήτηση για το πρασίνισμα. Κάποια καλλιέργειες πρωτεϊνούχων ε, φυτών μπορούν να εντάσσονται στην βιοπικιλότητα ε, για παράδειγμα το αλφα-αλφα είναι καταπληκτική καλλιέργεια που μπορεί να συμβάλλει στην βιοπικιλότητα και ούτως ή άλλως ε, δεν προϋποθέτει ισορές. Σε ό,τι αφορά τα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι οι γεωργοί μας χρειάζονται ένα είδος συμβολέου εμπιστοσύνης, αλλά και μία περίοδο προσαρμογής. Τι εννοώ με το συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Ε, υπάρχουν πολλά, πολλές απαγορεύσεις και έχουμε και ένα προηγούμενο με την οδηγία πλαίσιο για το είδωρ. Εκεί προβλέπονται κάποιοι στόχοι αποτελέσματος, αλλά όχι υποχρέωση συγκεκριμένου μέσου. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι γεωργοί είναι έξυπνοι άνθρωποι. Αν τους προτείνουμε λοιπόν στόχους προσιλοποίηση με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα θα δείξουν ευρηματικότητα και θα δείξουν την απαραίτητη δημιουργικότητα και με υπερηφάνεια θα επιτελέσουν το έργο τους ε, υλοποιώντας το στόχο. Και με τις τροπολογίες μας θα μπορούσαμε προς αυτή την κατεύθυνση να χαράξουμε ένα νέο δρόμο. Τις προάλλες είπα σε μια άλλη συζήτηση που έγινε σε ό,τι αφορά το θέμα της ανανέωσης του κεφαλαίου, του ανθρώπινου κεφαλαίου, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε ανησυχίες για την ικανότητα παραγωγής, για την αύξηση του πληθυσμού, έχουμε ε, προβληματισμό ως προς την αυτάρκεια την επιστημιστική. Αν όμως ε, δεν έχουμε αρκετούς ε, γεωργούς και αρκετές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ό,τι και να κάνουμε είναι περιττό. Το θέμα των νέων γεωργών είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να το λάβουν δεόντως υπόψη. Σε ορισμένες χώρες έχουμε μεγάλο ρυθμό μικρών καλλιεργειών. Εκεί το θέμα της ανανέωσης των γενεών δεν είναι άμεσο ούτε οξύ. Όταν βλέπουμε όμως τα στοιχεία ανακράτος και όταν βλέπουμε τις, ε, τις, ε, επιφάνειες, και το μέσο ηλικιακό όρο, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Και πολλές φορές ε, είναι κάπως κτητική Γιώργη, ε, αλλά ε, σίγουρα είναι πολύ σωστό ότι ένας αποκλεισμένος, απομονωμένος Γεωργός ε, είναι ένας Γεωργός που κινδυνεύει. Αυτό θα το πρέπει να το έχουμε υπόψη και πραγματικά χαράχτηκαν εξίδηλα στη μνήμη μου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό των ενεργών Γεωργών, συμφωνώ με τον εισηγητή να ορίσουμε, να θεσπίσουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινοτικό ενωσιακό πλαίσιο, αλλά μετά να και στη διακριτική ευχαίρεια του κράτους μέλους να το διευκρινίσει, να το συγκεκριμενοποιήσει. Ε, το θέμα της ε, οικοαιρεσιμότητας, ένα σημείο που δεν αναφέρθηκε. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η οικοαιρεσιμότητα στις διάφορες χώρες μας οδηγεί σε έναν ε, ανταγωνισμό που ε, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως αθέμητος υπό το πρίσμα της ενίας αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε καλύτερα, να συγκεκριμενοποιήσουμε καλύτερα τι περιμένουμε από την οικοαιρεσιμότητα. Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες επιφάνειες, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, επεκτείνει την ενίσχυση σε ανακτάριο σε όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε βέβαια την έκθεση Dorfman και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες διευκρινήσεις. Εγώ σας είπα ότι το να ανοίξουμε τα, τα ποιοτικά κρασιά στις α, ε, ε, πληρωμές ε, αναεκτάριο δεν είναι σωστό. Ε, γιατί μερικές φορές είναι σαν λιμοσύνη αυτό το θέμα των, ε, των ενίσχυσεων αναεκτάριο. Το ίδιο ισχύει για τα απορροκυπευτικά. Εγώ προτιμώ να έχουμε μία επιλεξιμότητα, αλλά όχι μία συστηματική επιλεξιμότητα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σαλβάμα. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Καπούλα Σάντον, διότι οι ιδέες του διέπονται από την, κοινωνική, από την κοινή λογική και μάλιστα επισκέφθηκε και τη Φιλανδία σε μια περίοδο που δεν ε, φυτρώνει τίποτα το Φεβρουάριο, άρα παρόλα αυτά ήταν καρποφόρα η συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να τα σχολιάσω και εγώ με τη σειρά που τα παρουσίασε ο κύριος Καπούλα Σάντος. Φυσικά δεν μπορεί να περιμένουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό ο οποίος θα ικανοποιεί κάθε κράτος μέλος αυτό το τόσο περίπλοκο ζήτημα. Αλλά για το θέμα του greening Έχω να κάνω κάποιες επισημάνσεις παρά το γεγονός ότι κάποια έχουν ήδη αναφερθεί. Το θέμα του 30%. Θα πρέπει να συμφωνήσω με την Ελίζα Μπεθκέστιγκερ εδώ. Θα είναι πολύ, πιο, πολύ εύκολο να το δεχτούμε και θα στείλουμε και αμφιλεγόμενο μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι αν μπορούμε να δώσουμε κίνητρα για να κάνουμε περισσότερα στον πρώτο πυλάνα, ε, ωραίο θα ήταν, δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό, αλλά μέχρι τούδε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά όπως είπαν ε, και η Ελίζα Μπεδιέγκλε και ο Πίτερ Γιάρ και συμφωνώ και εγώ να με ε, σε περιλάβουν ως μέλος της ομάδας όταν συζητάμε για το δεύτερο πυλώνα και το τι έχει γίνει μέχρι τούδε. Ε, υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει σε πολλά κράτη-μέλη και θα πρέπει και εδώ να δράσουμε με γνώμενα την κοινή λογική και πάλι. Με χαρά επίσης άκουσα ότι αυτή η επέτηση των τριών εκταρίων θα πρέπει να είναι περίπου 20. Ακόμα και 15 να έχουμε, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάποιες περιοχές της Ευρώπης όταν αναφερόμαστε σε περιβαλλοντικές ε, τιμές, ε, δεν είναι λογικό να ζητάμε αυτομάτως ε, τρία εκτάρια, διότι η φύση δεν το απαιτεί. Γιατί να το απαιτεί αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον, θα πρέπει να συμφωνήσω και με τον Τζιμ Νίκολσον εδώ. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο διεξοδικοί εδώ, διότι Εάν ε, αποστέλουμε μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε πιο απλούς κανόνες και κατόπιν τους παρουσιάζουμε κάτι στο οποίο η απλούστευση και μόνον περιπλέκει τα πράγματα, δεν είναι απλώς ένα ζήτημα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου, αποτελεί πρόβλημα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών της. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσέξουμε τι εννοούμε με τον όρο απλούστευση. Είναι σαν να παίρνει κάποιο ασφάλεια ζωή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να στέλνουμε ω μήνυμα στου Ευρωπαίου πολίτε ότι ε, η γεωργία είναι πολύ πιο ακριβή όταν υποτίθεται ότι ε, θέλουμε να είμαστε λιγότερο παραγωγικοί ω προ τη στήριξη. Ε, δεν είναι λογικό αυτό. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, η συνδεδεμένη στήριξη χρειάζεται πράγματι σε κάποιες χώρες, αλλά όπως είπε και η Μαρή, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και καλό θα ήταν να μας πούν και πώς ακριβώς θα είναι ο ορισμός όταν επιτρέπεται αυτή η εσωτερική σύγκληση μεταξύ πυλώνων. Κάποιος είπε μάλιστα ο κύριος Σάντος νομίζω το είπε, ότι αν είναι μόνο το 25% του δεύτερου πυλώνα, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο του 10% από τον άλλο πυλώνα. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και ο διάβολος, όπως γνωρίζουμε, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σε γενικές γραμμές όμως, εξαιρετική δουλειά κύριε Καπούλα Σάντος και σας ευχαριστώ. Κύριος Βοητσεχόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εξετάζουμε ένα από τα, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις, για να μην πω τι σημαντικότερη έκθεση αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί η έκθεση αυτή αφορά το σημαντικότερο τμήμα της σπουδαιότερης ε, κοινοτικής πολιτικής, την γεωρική πολιτική και το σημαντικότερο τμήμα της γεωρικής πολιτικής που είναι οι άμεσες πληρωμές. Θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμής προς τον εισηγητή και να εκφράσω την αναγνώριση και το θαυμασμό μου για το πολύ αξιόλογο έργο που επιτελεί. Και από πολλές συζητήσεις που είχαμε προσπάθησε να συνδυάσει τις διάφορες προτάσεις και είναι αξιοσέβαστη η προσπάθειά του να καταλήξει συμβιβασμούς. Βέβαια αυτό το διαλλακτικό πνεύμα έχει και κάποια όρια και τα όρια αυτά προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία, από την ενωσιακή νομοθεσία και για αυτά τα όρια πολύ λίγα λέμε. Η μεταρρύθμιση της κοινή ιωρικής πολιτικής δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα αλλά και νομικό ζήτημα, νομικό πρόβλημα. Έχουμε τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί εντοπίζονται πολύ σημαντικά προβλήματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν, να μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά. Το θέμα του, το θέμα του greening, του πρασινίσματος. Εγώ φυσικά είμαι υπέρ μιας γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό το στοιχείο του πρασινίσματος, αλλά δεν υπάρχουν βάσεις στη συνθήκη, νομικές βάσεις, για να επιβάλλουμε στους γεωργούς μας την υποχρέωση του πρασινίσματος. Δεν περιλαμβάνεται το πρασίνισμα στους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Άλλο ακόμη πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το θέμα της ανακατανομής των μέσων. Και εκεί σας παραπέμπω στη συνθήκη το άρθρο 18 για παράδειγμα, που απαγορεύει τη διάκριση λόγω α, εθνότητας. Ε, ε μετά τη μεταρρύθμιση η Λιθουανία, ο Λιθουανός Γεωργός θα λάβει ε, δύο φορές λιγότερες α, πληρωμές από ό,τι από την άλλη πλευρά της α, Ευρώπης. Γιατί? Για τους, ε, ε, για ποιους λόγους. Ε, μα για λόγους ε, συγκεκριμένης εκδοχής. Κάτι που απαγορεύει η συνθήκη. Στο άρθρο 32 της συνθήκης έχουμε τα όρια της ε, γεωργικής πολιτικής. Αναφέρθηκε εκεί, αναφέρεται εκεί η περιφερειακή διαφοροποίηση, όχι όμως η εθνική διαφοροποίηση. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δηλαδή οι διαφορές μεταξύ περιφερειών και όχι μεταξύ χωρών. Και τέλος, στο άρθρο 40 έχουμε σοβαρή απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σαφής και κατηγορηματική απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των γεωργών. Ως ε, Πολωνός Ευρωβουλευτής αισθάνομαι την υποχρέωση να τα επισημάνω όλα αυτά γιατί ε, το Πολωνικό Κοινοβούλιο πρόσφατα ε, υιοθέτησε ένα ψήφισμα αναφερόμενο, αναφερόμενο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και ζητώντας ε, την λήψη υπόψη των νομικών κολλημάτων και τον σεβασμό της συνθήκης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και έχω και συγκεκριμένη πρόταση και θα ήθελα να σας απευθύνω μια έκκληση. Θα ήθελα η Επιτροπή να εξετάσει την... και μάλιστα να διοργανώσει και δημόσια ακρόαση για τις νομικές πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Γιατί μιλούμε για πολλές και διάφορες πτυχές, για τις πολιτικές, τις οικονομικές πτυχές, αλλά φαίνεται ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τις νομικές πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ ή μάλλον ε, υπάρχει συμβατότητα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ με τη συνθήκη για την ε, εφαρμογή της, Ευρω... Ε, για την συνθήκη εφαρμογής εφαρμοστική συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις εδώ. Είναι σημαντικό η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να μην καταστρατηγεί σημαντικές νομικές διατάξεις της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τη γνώμη των νομομαθών για την διαλεύκανση όλων αυτών των σημείων. Γιατί θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι όταν εγκρίνουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή ε, ε, γεωργικής πολιτικής δεν θα παραβιάζουμε τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε κάποιες ε, αλλαγές στην ΚΑΠ εφόσον δεν έχει αποσαφινιστεί η συμβατότητα τους με τις ε, νομικές διατάξεις της συνθήκης. Παρακαλώ λοιπόν να, γίνει, να διοργανωθεί δημόσια κρόση για τις νομικές πτυχές των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα. Ε, από τη στιγμή που υποβάλλετε αυτή την πρόταση θα σας παρακαλούσα να την διατυπώσετε και γραπτός για να βοηθηθεί και η Γραμματεία και η Επιτροπή για να συγκεκριμενοποιηθεί ακριβώς ε, η πρότασή σας. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω ε, κάποια σύντομα σχόλια σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που θα επιδράσουν το επίπεδο των εισοδημάτων και το θέμα της, ε, των ενισχύσεων ανά εκτάριο. Και ένα άλλο πρόβλημα αφορά το κατά πόσο το greening αυτό, το πρασίνισμα, θα περιληφθεί στις ε, στοιχειώδεις διατάξεις και θα ήθελα να ζητήσω την άποψη του εισηγητού για τα θέματα αυτά και να του ζητήσω να μας κάνει κάποιες διευκρινήσεις και να μας στείλει και γραπτός φυσικά ε, τις παρατηρήσεις του. Γιατί πραγματικά είναι τόσο εκτενής ο κατάλογος αυτού των θεμάτων και είναι τόσο δύσκολα ορισμένα από αυτά, ώστε για να μπορέσουμε να αποφαθούμε υπέρ ή κατά των προτάσεων των εισηγητών, καλό θα ήταν να έχουμε και ένα κείμενο για να στηριχθούμε. Σας θέλω παρακαλώ λοιπόν κύριε εισηγητά να μας στείλετε γραπτός μία σύνοψη, αν μπορείτε, της σημερινής συζήτησης με όλα τα επιμέρους σημεία για να μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι πολύ λακωνικός γιατί έχουμε και άλλο πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις αλλά πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω για το εξαιρετικά επικοδομητικό πνεύμα που πριτάνευσε στην απογευματινή συζήτηση και ελπίζω αυτό το πνεύμα να μας χαρακτηρίσει καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων και για όλα τα σημεία Διαπιστώνω πάντω ότι όλοι οι συνάδελφοι και όλε οι πολιτικέ παρατάξει ενστερνίζονται αυτό το πνεύμα συνεργασία και συμμερίζονται την ανάγκη ανέβρεση λύσεων για τα θέματα που μα ε, υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να έχουμε στεναρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να είναι ισχυρή και η διαπραγματευτική μα θέση απέναντι στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ελάχιστο χρόνο διαθέτουμε ακόμη, οπότε οι εισηγητές δεσμευθήκαμε μέχρι τα μέσα του Μαΐου να υποβάλουμε για μετάφραση γραπτό στην έκθεσή μας, ώστε να μπορέσουμε να Έχουμε όλες τις μεταφράσεις τον Ιούνιο, να γίνει η παρουσίαση 18 και 19, δεν κάνω λάθος, των διαφόρων επιμέρους εκθέσεων για τη γεωρική πολιτική. Ουσιαστικά δηλαδή έχω μόνο τρεις εβδομάδες στη διάθεσή μου για ένα τιτάνιο έργο της διαμόρφωσης ε, της έκθεσης. Οπότε παρακαλώ τους συναδέλφους, όσους έχουν προτάσεις που θέλουν να συμπεριληφθούν στην έκθεση, σας θέρμο παρακαλώ να μου τις στείλετε το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση αυτή την εβδομάδα. Επίσης ε, είμαι ανα πάση στιγμή στη διάθεσή σας, όπως έκανα και μέχρι τώρα, και πρόθυμος για διμερείς επαφές, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα περίπλοκα που είναι δύσκολο να τα εξηγήσουμε εδώ. Σήμερα ε, διαπίστωσα ότι μερικοί συνάδελφοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη τι σημαίνει greening, τι σημαίνει πρασίνισμα ή το θέμα της διπλής ε, πληρωμής. Ένα ζήτημα που προβλημάτισε πολλούς συναδέλφους. Για το θέμα της διπλής πληρωμής δεν είδα κανένα να ενδιαφέρεται και να προβληματίζεται όταν υπάρχουν σήμερα άμεσες πληρωμές στον πρώτο πυλώνα και πληρωμές για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα για την ίδια ακριβώς γεωρική έκταση. Αυτό κανένα πρόβλημα δεν δημιούργησε. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ή δεν επισήμανε νομικό κόλλημα. Είναι μια πρακτική που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιες ε, και τεχνικές και νομικές αλλά και δεοντολογικές λύσεις όπως είναι προφανές ότι χρειάζονται. Δεν χρειάζεται τώρα να ανατρέξουμε όλες τις παρατηρήσεις ε, και τις προτάσεις. Επιβεβαιώθηκαν πολλές ανησυχίες ε, και αμφιβολίες μου. Θέλουμε φυσικά να βρούμε κάποιες τεχνικές λύσεις, πάντως νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ως προς το πρωταρχικό ζήτημα που είναι η αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης και η διαπραγματευτική μας στρατηγική. Ως προς αυτό νομίζω υπάρχει ε, διακομματική συμφωνία. Πιστεύω ότι κατάλαβα το βασικό, τους βασικούς προβληματισμούς και θα προσπαθήσω να τους συμπεριλάβω στην έκθεση που θα συντάξω στο εγγύς μέλλον. Δεν θέλω τώρα ούτε προλαβαίνω να απαντήσω διεξοδικά σε όλες τις παρατηρήσεις σας. Πάντως θα αναφερθώ στα τελευταία σχόλια του Προέδρου. Αν κατάλαβα καλά, μίλησε για, τις, για τη σημασία που έχουν οι άμεσες πληρωμές στο εισόδημα των γεωργών. Σε μια ανταγωνιστική, ανοιχτή στον ανταγωνισμό γεωργίας στην Ευρώπη, που μερικές φορές είναι και αθέμητος ανταγωνισμός, χωρίς άμεσες πληρωμές, πολλές βασικές ε, δραστηριότητες ε, που είναι απαραίτητες για μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή γεωργία δεν θα ήταν ε, ε, δυνατή. Μια τέτοια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή γεωργία δεν θα ήταν δυνατή σήμερα χωρίς άμεσες πληρωμές. Σε ό,τι αφορά τη βασική πληρωμή, για την οποία επίσης εκφράστηκαν πολλές αμφιβολίες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε βασική πληρωμή αν δεν προσδιορίσουμε προηγουμένως τους κανόνες και τα κριτήρια πρόσβασης σε αυτή την πληρωμή. Ας μην τα μπερδεύουμε. Υπάρχει μια βασική πληρωμή και απαιτείται εδώ η Οπότε θα πρέπει να ε, αν έχουμε μια πληρωμή greening που ε, προϋποθέτει επιπλέον κριτήρια και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να λάβει ο Γεωργός την ενίσχυση. Θα βρούμε πάντως πιστεύω λύση. Ο κύριος Βοητσεχόφσκι Αχ, είναι πολύ δύσκολο το όνομά σα, ε, κύριε Βοητσεχόφσκι. Αυτά τα πολωνικά ονόματα είναι δύσκολα στην προφορά. Εν πάση περιπτώσει, μίλησε για ζητήματα πολύ πιο θεμελιώδη που ξεπερνούν τη σημερινή συζήτηση. Είναι τα νομικά ζητήματα, οι νομικέ πτυχέ. Πιστεύω όμω ότι για τα θέματα αυτά τα νομικά, οι υπηρεσίε μα και η, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσουν δημόσιε ακροάσει ώστε να διασκεδαστούν οποιασδήποτε αμφιβολίε για την ε, για, το, για την νομιμότητα ε, ή τη συμβατότητα των διατάξεων αυτών με την συνθήκη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωση ή τη συνθήκη της Λισαβόνας. Φυσικά θα πρέπει να διασκεδαστούν οποιασδήποτε αμφιβολίες που υπάρχουν για την νομιμότητα των διατάξεων που θα κληθούμε να εγκρίνουμε. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Είμαι πρόθυμος, είμαι στη διάθεσή σας και διμερός να το συζητήσουμε, να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίες σας ακόμη και στα διαλύματα μεταξύ των συνεδριάσεων και στείλτε μου τις προτάσεις σας το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, πολύ πιθανό και μετά τον Ιούνιο να έχουμε μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων με υποβολή τριοπολογιών, με διαμόρφωση συμβαστικών πρωτοβουλειών, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια μεστή και συνενετική στεναρή πρόταση που θα ενισχύσει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις και θα διατρανώσει το ρόλο μας ως συνομοθέτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ε, επίσης, ε, για να διευκολύνουμε και τον εισηγητή μας και να μπορέσει να διαμορφώσει εγκαίρως την έκθεσή του, θα στείλουμε το συντομότερο δυνατό τις προτάσεις μας. Γιατί και μας μας ενδιαφέρει να είναι καλή έκθεση του εισηγητού. Παρακαλώ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι δυνατός, το συντομότερο δυνατό γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και νομίζω ότι κύριε Καπούλα Σάντος δώσατε μία πρώτη εντύπωση για το πώς θα διαμορφωθεί η έκθεσή σας και εγώ συμφωνώ με πολλούς γερμανόφωνους ότι σε κάποια σημεία δεν κατάλαβα ε, ακριβώς τι θα περιλαμβάνονται ε, στις λεπτομέρειες αλλά αυτό θα ευκρινίσουμε κάποια σημεία τώρα στα οποία έχω παρτρήσει να κάνω σε ό,τι αφορά τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση η οποία βασίζεται αφενός σε μια προσέγγιση των επιπέδων ε, στήριξης ε, μεταξύ κρατών μελών και αφετέρου ε, τη συμπερίληψη και άλλων παραγόντων τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία έλαβα τα έλαβα, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξα, αλλά φυσικά θα πρέπει να δούμε το σύνολο του σχεδίου σας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκφέρουμε άποψη σε, από αυτόν. Πολύ σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση ήταν ο παράγοντας του greening. Ένα θέμα ήταν η διάκριση μεταξύ των βασικών πληρωμών και του greening. Κοιτώντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντως πρόκειται για δύο ξεχωριστές πληρωμές. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν ληφθεί αυτά υπόψη, αυτά που αποτυπώνται στη συζήτηση. Ένα άλλο θέμα είναι οι κυρώσει οι οποίε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπέβαλε σχετικό έγγραφο εργασίας, το οποίο ήταν προ τα κράτη-μέλη, αλλά το έλαβε φυσικά και το Κοινοβούλιο, όπου παρουσιάσαμε μια αναρακτική λύση, η οποία τη λέει ότι φυσικά δεν έχει, δεν υπάρχει επίπτωση ε, σε ό,τι αφορά το greening, σε ό,τι αφορά τις βασικές πληρωμές, αλλά αν κάποιος δεν συμμετέχει καθόλου στο greening, ε, ίσως ε, οι κυρώσεις θα πρέπει να ξεπερνούν το 30%. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο στην αγροτική πολιτική, το ξέρουμε και από προηγούμενα μέτρα για την αγρανάπαυση και το καθεξής. Η κύρωση που ξεπερνά το 30% δηλαδή δεν ε, αποτελεί όμως άμεσα μείωση του βασικού ποσού Στη συνέχεια, μιλήσατε για ενδεχόμενο ελάχιστο όριο 20 εκταρίων για την ε, διαφοροποίηση. Εγώ είχα καταλάβει ότι αυτό ε, θα ίσχυε βασικά για τις ε, επιφάνειες οικολογικής εστίασης. Μας φαίνεται πάρα πολύ υψηλό αυτό το αυτές οι εκτάσεις. Γιατί έτσι αποκλείονται και ολόκληρα κρατημέλη. Νομίζω ότι θα δυσκόλευε το greening πάρα πολύ. Εμείς είχαμε προτείνει όριο τριών εκτάριων για την διαφοροποίηση. Γιατί αλλιώς την νόημα έχει η ελάχιστη έκταση σε ό,τι αφορά τα συστήματα εκπεριτροπής για το greening προσπαθήσαμε να βρούμε μία λύση η οποία ε, συνάδει με την αρχή της ετήσιας πληρωμής. Αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τους ε, ελέγχους και θα ήταν κατά του γενικότερου στόχου της απλούστευσης για την καλλιέργεια συγκεκριμένων ε, φυτών, θεωρώ ότι αυτό θα παρουσίαζε προβλήματα και σε ό,τι αφορά τον greening αλλά και σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ. Natura 2000, το ακούσαμε, που δεν συμπεριληφθήκε στο greening για τον απλό λόγο ότι το πρόγραμμα Natura 2000 δεν συνεπάγεται ουσιαστικά επιπλέον υποχρεώσεις για τον γεωργό, αλλά ουσιαστικά ε, χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν μεμονωμένα σχέδια εκμετάλλευσης των εκτάσεων αυτών. Αυτό δεν ισχύει δυστυχώς παντού. Σε ό,τι αφορά τον ενεργό γεωργό τώρα. Αναφέρθηκε ότι είναι υπερβολικά περίπλοκο το σύστημα αυτό και ότι θα, συνε... θα σήμαινε μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. Εξετάζουμε ένα μοντέλο στην παρούσα φάση το οποίο θα βασιζόταν σε έναν αρνητικό κατάλογο κάποιων δραστηριοτήτων τις οποίες δεν ε, συμπεριλαμβάνουμε στις άμεσες πληρωμές, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί απόλυτο λόγο εξαίρεσης και αποκλεισμού. Απλά επαφίεται στις ε, εκάστοτε επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι είναι όντως ενεργή γεωργή, για να αποφύγουμε ενδεχόμενους, ε, ενδεχόμενες περιπτώσεις αρνητικής διάκρισης. Για να μην υπάρχει δηλαδή ε, πρόβλημα διακριτικής μεταχείρισης κάποιων επιχειρήσεων. Αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης ουσιαστικά. Και αυτό θα είχε το πλεονέκτημα ότι θα μειώνονταν δραστικά ο αριθμός των ε, σχετικών επιχειρήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κάπινγκ και το greening, ακούστηκαν δύο ιδέες. να συμπεριληφθεί ένα ποσό καινοτομία ή να συμπεριληφθούν οι βασικές εκτάσεις. Στο greening, στο πρασίνισμα, αναφέρθηκε ενδεχομένως μεταφορά των ε, μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων στο δεύτερο πυλώνα. Θεωρώ ότι και οι δύο προτάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν γραφειοκρατικά. Θα σημαίνουν μεγάλη περιπλοκή των ζητημάτων αυτών. Δεν θα είχαμε μόνο το κόστος του εργατικού δυναμικού, αλλά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη και, άλλες, ε, και άλλα μέτρα και άλλα ποσά τα οποία είναι δύσκολα μετρήσιμα. Και για τη μεταφορά ε, μέσων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, αυτό θα σημαίνει ότι θα, πρέπει να, θα έπρεπε να προσαρμόζουμε κάθε χρόνο τα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφήστε που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε πότε ακριβώς ε, δεν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά. Και δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε τον προγραμματισμό του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για τέτοια σχετικά μικρά ποσά. Γενικά, στο, υπό το πρίσμα της απλοποίησης, της απλούστευσης, σε ό,τι αφορά το 15% ε, διοικητικά κόστος. Πρόκειται για έναν αριθμό ο οποίος προήλθε από την ε, μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν αναφέρεται στην όλη μεταρρύθμιση, αλλά μόνο στις άμεσες πληρωμές. Αναφέρεται, μάλλον δεν συμπεριλαμβάνει ένα παράγοντα, τον οποίο θα ήθελα να τονίσω, την πρότασή μας προκειμένου στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν καλά συστήματα ελέγχου που λειτουργούν σωστά, να έχουν τα κράτη-μέλη αυτά τη δυνατότητα να μειώσουν αυτά τα ποσοστά για τον έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού. Και θα σήμερα σημαντική απλούστευση ε, στα κρατη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το στοιχείο αυτό. Νομίζω ότι κοιτώντας αν κοιτούσαμε τι ισχύει για όλες τις χώρες, δεν θα καταλήγαμε στο 15% αλλά σε πολύ, διαφορετικές, σε πολύ διαφορετικά νούμερα. Πρώτο τελευταίο ζήτημα για τις πράξεις καταξιοδότησης. Οι πράξεις καταξιοδότηση ε, κατοχυρώνονται νομικά και νομίζω ότι αυτό είναι καλό γιατί έτσι εξασφαλίζεται ευελιξία και παράλληλα εμ, διασφαλίζεται ο πρωταγωνιστικός ο ρόλος στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει να το συζητήσετε με τα κρατημέλη γιατί από εκεί προέρχεται η βασική αντίσταση. Τελευταίο ζήτημα. Την πρότασή μας την ελέγξαμε και νομικά ασφαλώς, ενδελεχώς και σας διαβεβαιώνω ότι η πρόταση όπως κρατέθηκε στέκει νομικά. Και κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί ότι θα προσαχθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω ακριβώς του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα, γι' αυτό και δεν στερήσαμε από κανένα, ότι περιορίσαμε το λόγο, το χρόνο αγόρευσης. Τώρα, οργανωτικά, Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα που πολλές φορές φοβίζουν και πώς θα πρέπει για τα θέματα αυτά να αντιμετωπίσουμε, πώς θα μιλήσουμε με τους γεωργούς. Είχαμε τις εκθέσεις Χέρτσεκ, Ντες, Σάντος. Φαίνεται ότι βαίνουμε προς μια κατεύθυνση απλούστευσης, ότι θα είναι όλα πιο εύκολα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια περιπλοκή, μια τέτοια δυσκολία. Είναι τόσο δυσανάγνωστα πολλές φορές αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά πώς θα τα εξηγήσουμε στους γεωργούς μας. Και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά και πού θα μας οδηγήσουν όλα αυτά. Θα ήθελα να πω εν κατακλείδη ότι η έκθεση του κυρίου Βοητσεχόφς και αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση τελών Μαΐου ή αρχών Ιουνίου ε, και ίσως ε, θα πρέπει να προβλέψουμε νέα ημερομηνία για την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το μελλοντικό κριτήριο για τον καθορισμό των μειονεκτουσών περιοχών. Δυστυχώ δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Θα πρέπει να το κανονίσει η γραμματεία μα με του εκπροσώπου τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Δυστυχώ δεν προλάβαμε σήμερα να εξετάσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, γιατί δεν μα μας έφτασε ο χρόνο έπρεπε να ασχοληθούμε διεξοδικά με το πολύ σημαντικό θέμα των άμεσων πληρωμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. Α, συγγνώμη, κυρία εισηγητρία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω το, ε, να συμπεριλάβετε στην ενημερήσια διάταξη την ε, ημερομηνία για την συζήτηση αυτή, γιατί σε ένα κράτος μέλος γίνεται μία συζήτηση για το δεύτερο πυλώνα και θα πρέπει τέλος να γνωρίζουμε τι είναι η περιοχή. Για όλα, μάλλον όλα αυτά ε, μου είναι ακόμα πολύ περίεργα. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλήσω να προβλέψετε και επαρκή χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Μισή ώρα μου φαίνεται πάρα πολύ λίγη. Ε, τουλάχιστον μία ώρα, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα, πολύ ανοιχτά, πάρα πολλά ανοιχτά ερωτήματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Και το συντομότερο δυνατόν, παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κύριος Νίκολσον, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο που έθεσε το θέμα αυτό. Πολλές φορές έχω μείνει εδώ, όχι γιατί δεν ήταν εξαιρετική συζήτηση που κάναμε, αλλά και γιατί περίμενα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσω ε, κάτι άλλο. Γιατί... για τις μειονεκτούσες περιοχές. Είναι πάρα πολύ αυτοί που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε οργανώσει κατάλληλο χρόνο συζήτηση, να ξέρουμε πότε θα είναι η συζήτηση. Ε, και να γίνει όπως πρέπει. Υπάρχει χρόνος αύριο το πρωί γιατί η έκθεσή μου που πρόκειται να ψηφιστεί αναβάλλεται και επομένω αυτό σημαίνει ότι έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Δεν θα πω εγώ στη γραμματεία τι να κάνει και πώς θα οργανώσει την ημερήσια διάταξη διότι εγώ δεν τολμώ καν να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά θα ήθελα να είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει να συζητηθεί σε ώρα που μπορούν να είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής γιατί είναι σημαντικό. Και ε, αφού είναι εδώ πρόσωπο της Επιτροπής θα ήθελα να του πω κάτι. Λέει ότι το 15% είναι αυτό που είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι πολύ μεγάλο. Το 20% είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι υψηλότερο, χαμηλότερο. Ποιο είναι το σωστό ποσοστό. Μήπως πρέπει να ε, δει την πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας πει ποιο είναι το πραγματικό κόστος ε, της διαχείρισης ε, των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να πληρώσουν τα κράτη-μέλη για να διαχειριστούν τις προτάσεις τους. Ε, λυπούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Θα πρέπει να το βάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να, απαντήσουν, να απαντήσει γραπτός. Ένα λεπτό μας έχει μείνει ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους δύο προηγούμενους ομιλητές. Είναι περίεργη η κατάσταση γιατί εδώ και καιρό περιμένουμε αυτή τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την προηγούμενη εβδομάδα ε, Είχαμε υποβάλει και ένα ερώτημα προς το Συμβούλιο στην Ολομέλεια, το οποίο ε, απαντήθηκε χωρίς σεβασμό και χωρίς ικανοποιητικό τρόπο. Ε, ήταν πραγματικά παράδειγμα ο τρόπος που ε, συμπεριφέρθηκε το Συμβούλιο, παρουσιάστηκε αργά, δεν απάντησε σωστά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να έχουμε χρόνο προκειμένου την επόμενη φορά να μην βρεθούμε πάλι υπό χρονική πίεση. Ναι. Παρακαλώ να ενημερώσει η Γραμματεία για τις παρατηρήσεις του κ. Ντόρφμαν τον πρόεδρο Δεκάστρο και να το θέσουμε και στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε την επόμενη φορά να προβλέψουμε περισσότερο χρόνο και για την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Λυπούμε στο συγγνώμη από τους διερμηνείς για τη μικρή παράταση του αερίου. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεδρίαση. Καλό απόγευμα.